Έχουμε μια πολύ υπερφορτωμένη ημερήσια διάταξη μπροστά μας και δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Eh, λοιπόν, εντάξει, ελπίζω ότι έχετε τις κάρτες μαζί σας για να ψηφίσουμε, να ψηφίσετε. Ε, δεν έχετε, τι γίνεται. Ζητήστε, και από τον βοηθό να ζητήσετε να την φέρει, εγώ την έφερα τη δική μου, εντάξει γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες μπροστά μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον τουριστικό προορισμό, πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο η Ευρώπη. Έχουμε 57 τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι η κυρία Ρόνερ θέλει να παρέμβει. Θέλετε να παρέμβετε? Όχι. Περνάμε άμεσα στην ψηφοφορία λοιπόν. Πολύ ωραία. Παράγραφος 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ μια στιγμή ξεχωριστή σε τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ τι είπατε αποσύρθηκε το είδανε Ζητώ συγγνώμη, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. Προφορική τροπολογία 2. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 19. Μανέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά επαναλαμβάνουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 30 από την άλλη σελίδα την άλλη πλευρά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 και 54 είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 39 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε μάλιστα ο, ο λίστημα 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 44 αποσύρθηκε προφορική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 55 52 διορθώνει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία με την κάρτα σας αν την έχετε αλλιώς θα προσμετρήσουμε μετά αρχίζει η ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ναι ναι εντάξει Έχουμε λοιπόν 22 υπέρ, α, άλλος ένας 24 υπέρ, καμία ψήφος εναντίον, 25 υπέρ και κανείς εναντίον. Εξαιρετικά. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ ως εισηγήτρια θερμά για την έγκριση. Χαίρομαι πολύ για την τουριστική πολιτική που θα ακολουθηθεί και σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, περνάμε στη συνέχεια στο επόμενο σημείο. Ευρωπαϊκό έτος ε, ε δραστήριας γύρανσης. Ο Χάνο είναι υπεύθυνο. Έχεις να πεις κάτι Χάνο Τάκουλα. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου που δεν έχεις να πεις και τίποτα. Ευχαριστώ. Και περνάμε στην ψήφιση τώρα, στην ψηφοφορία. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Και πάλι επαναλαμβάνουμε. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αποτέλεσμα. 12 υπέρ, 14 εναντίον. Απορρίφθηκε. 14 εναντίον. 12 υπέρ. Απορρίφθηκε. Θέλατε να ψηφίσετε πώς εσείς, τι θα ψηφίζατε. Εντάξει, και πάλι λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 7. Όσοι είναι λοιπόν υπέρ, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 13 εναντίον. Και ο Χάνο, εσύ είσαι κατά. Χάνο. 14-14. Ισοψηφία απορρίπτεται. Μάλιστα. It Καταπίπτει λέτε, εντάξει, ωραία, έγινε. Ωραία. Χάνω. Φέρε την κάρτα σου για να συμμετέχει στην ψηφοφορία. Βε την κάρτα σου, εντάξει. Amendment 8. Υπολογία 8, υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 10. Λίγη η ψηφοφορία. Ισοψηφία 14-14 απορρίπτεται. Α, και εσύ χάνω. Ωραία, έστω λοιπόν, απορρίφθηκε. Ωραία, τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 13 υπέρ 14 εναντίον απορρίφθηκε. Χάνω ήσουν και εσύ εναντίον. 13 υπέρ 15 εναντίον. Πολύ ωραία. Έχει ιδιαίτερη μεταχείριση σήμερα, τη οποία την χάνει εδώ. Πού πάμε μετά στην τροπολογία 13. 13 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14. Τι λες? Πρέπει απλά να επανέλθουμε στην 12. Ξανά η 12. Υπέρ. Σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται αυτό το δεύτερο τμήμα. Και η τροπολογία 1 του εισηγητή υπέρ. Εντάξει, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 1. 13 την καλύψαμε. Ναι, καλύφθη. Πάει αυτή. 14 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 2. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 15 Ήδη καλύπτεται από την τροπολογία 2 ή όχι. Να ψηφίσουμε. Εντάξει. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 15. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 16 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 17 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε τη 17 πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 17 υπέρ 12 εναντίον εγκρίνεται η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 19 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 19 πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 27 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα εγκρίνεται 27 εγκρίνεται 28 τώρα υπέρ κατά εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά Α, θα ελέγξουμε ε, περνάμε στην 31 απορρίφθηκε 29 υπέρ κατά αποχές άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 31 πέρας ψηφοφορίας Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 38 πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε με ισοψηφία 15-15 εντάξει προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 43 εντάξει 43 όχι 40 όχι εντάξει 43 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ ποια λέτε εσείς η 43. Εντάξει, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τη 43 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ. Μάλιστα. Ε, σαφές το αποτέλεσμα. Υπεψηφίστηκε Η 45 υπέρ. Συγγνώμη, μια στιγμή. Ε, δημιουργήθηκε μια σύγχυση εδώ. Η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 6, μόνο η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα, 29 υπέρ, κανείς εναντίον. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια Χάνο Τάκουλα. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Τάκουλα. Πρόεδρος, εντάξει. Λοιπόν, περνάμε τώρα... Αν μπορώ να μιλήσω και γερμανικά, εντάξει. Είναι τόσο κουραστικό να μιλάει κανείς πάντα αγγλικά. Θα μιλήσω τώρα γερμανικά. Αν θέλετε να με καταλάβετε, φορέστε ακουστικά. Λοιπόν, προς χαρά μεγάλη των διερμηνέων, λέει η Πρόεδρος. Πάλι του Χάνο είναι αυτό το θέμα. Μα τι γίνεται εδώ. Ε, τώρα φτάνει πια Χάνο, εντάξει. Ε, επήλθε ο κόρος. Ναι, πάλι, πάλι έκθεση. Και πώς γίνεται αυτό, έτσι. Λοιπόν, η κοινωνική ένταξη των Ρωμά, των συγκάνων. Αυτό είναι το θέμα που θα ψηφίσουμε. Ναι, παρακαλώ, εσείς. Αντίθετα από αυτό που αναφέρεται στο έγγραφο, δεν ε, προσυπογράφουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Εντάξει δεν υποστηρίζετε την ε, συμβαστική τροπολογία 3, έτσι. Ωραία. Ε, τώρα πια γερμανικά πάλι. Λοιπόν, η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 1, ψηφίζουμε. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Εσείς είσαστε εναντίον. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, εγκρίθηκε. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Σημείο 2 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 3. Υπέρ. Συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 4. Πέρας ψηφοφορία. Λοιπόν, εγκρίθηκε 23 υπέρ, 8 εναντίον. Συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά, Αποχέ. εγκρίθηκε. Η τροπολογία 8 υπέρ. 8 κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 10 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 10. Πέρας ψηφοφορίας, αποτέλεσμα 18-13, <clears throat> εγκρίθηκε. Συμβασμός 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το πρώτο. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το δεύτερο. 16 υπέρ κατά διορθώνεται 18 λέγεται στην πρόεδρο. Η 16 τι είναι καταπίπτει. Α, είναι μέρος του συμβιβασμού λέτε. Εντάξει, πολύ καλά. Εντάξει. Και η 17 επίση πολύ καλά. Δεν ήταν απόλυτα σαφές, αλλά έστω. Η 18 τώρα, Μαρία Μπαντία Κουτσέτ, υπέρ τη 18, κατά. απόχέ εγκρίθηκε. Η 19 υπέρ, κατά. απόχέ εγκρίθηκε. Η 20 υπέρ, κατά. απόχέ εγκρίθηκε. Η 21 υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίθηκε. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε που πάμε τώρα 25 25 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά εντάξει άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 29 καβαντά πέρας ψηφοφορίας ε, πολύ μικρή διαφορά 16 υπέρ 15 εναντίον εγκρίθηκε η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 32 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 32 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 36 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίθηκε. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 49 και 51 είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Προφορική τροπολογία 2. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 54. Όχι, όχι. Α, εντάξει, 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 59 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την 59, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, πέρα ψηφοφορία είπα. Το προσέξατε. Τι γίνεται με τις οθόνες. Α, ένας παραπάνω. Α, ούτως ή άλλως. Εντάξει, οκ. Αποτέλεσμα. 11 υπέρ 19 εναντίον. Απορρίφθηκε. 11-19. Βερονίκ, με, να καταμετρήσει να δεις ο αριθμός να είναι ο σωστός. Να μην υπάρχει ένας παραπάνω. 11-19. Απορρίφθηκε λοιπόν. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 67 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 71 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 71 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 17-13 εγκρίθηκε συγγνώμη 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Πέρας ψηφοφορίας. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα παραπάνω. Πέρα, πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ. 2 αποχές. Μου είχαν πει ότι υπάρχει ένα μέλος παραπάνω του ΕΛΚ που συμμετείχε στην ψηφοφορία. Είμαστε πιο πολλοί, είμαστε τόσοι πολλοί παρόντες και είναι ένας παραπάνω. και εμού συμπεριλαμβανομένης 15 υπερβολικό αριθμό. πολύ μεγάλο. Χάνο. Τάκουλα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΛΚΑ για την υποστήριξή του. Είναι τόσο ενθουσιώδες οι βουλευτές για την έκθεση αυτή που ψηφίζουν περισσότεροι από όσοι, <laughs> πρέπει. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ και τους κοιόδους συζητητές. Ευχαριστώ όλα τα άτομα τα οποία με βοήθησαν για να δουλέψω επ' αυτών των δύο εκθέσεων. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ επίσης και τη Γραμματεία της Επιτροπής. Ευχαριστώ όλους τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Υπήρχαν κάποια μείον στον κατάλογο ψηφοφορίας. Προσπάθησα όμως οι τροπολογίες να είναι σύντομες και να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια πολλές φορές. Το βασικό ήταν να αποφύγουμε τις επαναλήψεις, ούτως ώστε αυτοί που διαβάζουν αυτές τις εκθέσεις να καταλαβαίνουν τέλος πάντων τι θέλουμε να πούμε. Φυσικά ο καθένας θέλει τη δική του φράση ας πούμε μέσα, αλλά πρέπει να αποφύγουμε τις επαναλήψεις. Στη Φιλανδία λέμε ότι αρκεί να πούμε κάτι μια φορά ξεκάθαρα και αρκεί. Αν ρωτήσω ας πούμε μ' και πω ε, ναι, σ' αγαπώ, αρκεί. Είναι, είναι ξεκάθαρο. Ενώ αν με ρωτήσει κάποιο με αγαπά και του πω ναι, ναι, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, σ' αγαπώ, δεν θα με πιστέψει τελικά. Γι' αυτό μερικέ φορέ οι επαναλήψει δεν είναι πιστικέ. Σα ευχαριστώ όλου και καλή συνέχεια για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Πρόεδρος, τώρα πάμε στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Κυρία Μπαντία Κουτσέτ, θέλετε τον λόγο παρακαλώ. Ναι. Απλά και μόνο να ευχαριστήσω μόνο για όλες τις παρεμβάσεις. Είχαμε 57 τροπολογίες που μεταφράστηκαν σε 6 συμβαστικές τροπολογίες. Επίσης να πω ότι κάποιες από τις τροπολογίες δεν μπορέσαμε να τις ενσωματώσουμε. Ήταν τροπολογίες επί των συμβιβασμών. Ήταν πολύ δύσκολο λοιπόν να ενσωματωθούν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ λοιπόν για τις προτάσεις. Και υποθέτω ότι έχουν καταμετρηθεί οι του ΕΛΚ και ξέρουν ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι όχι στην ψηφοφορία, εντάξει. Φυσικά γνωρίζουμε ποιοι πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, υπάρχουν εδώ και τα αναπληρωματικά μέλη, απλώς ε, συμμετέχουν χωρίς να ψηφίζουν βέβαια. Απλώς Απλώς παρακολουθούν, έτσι. Οι αναπληρωτές μου δεν συμμετέχουν. Απλώς είμαστε τόσο πολύ άριθμη ομάδα που έτσι μας αρέσει να συμμετέχουμε. Λοιπόν, η μηχανή είναι έντιμη και κέραια. Είπε η συσκευή είχαν ψηφίσει 1,5 παραπάνω. Αν εδώ έχουμε 15-3 δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν, ένα είχε ψηφίσει παραπάνω ούτω ή άλλω. Λοιπόν, να είσαστε προσεκτικοί εσεί οι τρει, να μην συμμετέχετε. Μάτουλα, ποιο άλλο, Μπέλετ και η κυρία και εκείνη όχι. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να συμμετέχουν. Περνάμε στην έκθεση. Συμβασμό 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 υπέρ. Την, η 8 λέγεται. Ναι, η 8, συγγνώμη. 8 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 9, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την, την 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αποτέλεσμα 24 υπέρ, 8 εναντίον εγκρίθηκε. Πολύ ωραία. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 11 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 11 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας πέρας ναι εγκρίθηκε 18 υπέρ 14 εναντίον η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 ναι 22 υπέρ κατά αποχές 22 μου είπαν. Αυτό μου είπαν. Λοιπόν, έστω. Ποιοι είναι υπέρ. 22. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 έχει αποσυρθεί αυτή συμβασμός 4 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περίεργο. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε, συγγνώμη, συγγνώμη, απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 53 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 30 υπέρ, δύο αποχές, καμία ψήφος εναντίον. Θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Μπάντια Ικουτσέτ. Ivan, παρακαλώ. Νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας σε 10 λεπτά, διότι υπάρχουν αυτά, υπάρχει αυτός ο χρόνος, θα είμαστε ελεύθεροι όμως στις 5 που έχουμε να συνεχίσουμε. Α, η κυρία Ρέντινγκ είναι παρούσα. Ήβαν, δεν γίνεται. Εντάξει, είναι εδώ η κυρία Ρέντινγκ. Ωραία, <laughs> σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Χαιρετίζουμε και καλωσορίζουμε άμεσα την Επίτροπο.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 Έχουμε και την απόφαση των συντονιστών. Τη λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τη χθεσινοβραδινή απόφαση των συντονιστών. Εάν θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να το πείτε τώρα. Δεν θέλω να εκφράσω κάποια αντίρρηση, αλλά θα ήθελα να έχω την πληροφορία για τα βραβεία Λουξ. Όταν γίνεται μετά από την παρουσίαση της Επιτρόπου να μάθουμε ποιοι πήραν τα βραβεία Λουξ. Αγαπητή κυρία Ρέντινγκ, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, χαρούμενοι που είσαστε παρούσα εδώ. Είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε πολλά θέματα που απομένουν από πέρυσι και θέλουμε φυσικά να γνωρίζουμε πώ εφέτο, τι θα κάνετε, πώ θα αντιμετωπίσετε τι διαφορετικέ δυνατότητε τη επικοινωνία όσον αφορά το έτος εθελοντών. Έχουμε και τα επόμενα δύο έτη τα οποία εξετάζονται για διαφορετικές διάφορες δράσεις. Θα λέγα ότι έχετε εξοικειωθεί και έχετε τόσο πολύ εργαστεί για αυτόν τον τομέα που μπορείτε με εξαιρετικό τρόπο να μας πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας. Ίσως και πιο εξειδικευμένη περιγραφή της αποκαλούμενης στρατηγικής. Ξέρετε ότι συμφωνώ μαζί σας στρατηγική ω όρο για τα θέματα επικοινωνία είναι κάπω δυσχερή. Αλλά τέλο πάντων έτσι αναφερόμαστε σε αυτό ω στρατηγική. Χαιρόμαστε γι' αυτό ώστε να υπάρξει, να προαχθεί αυτό το θέμα, να μπορέσουμε πιο διεξοδικά να το εξετάσουμε και να το δούμε αυτό το θέμα. Προσδοκούμε να ακούσουμε τι νέε σα ιδέε όσον αφορά τα θέματα ηθαγένεια, των πολιτών δηλαδή και τη επικοινωνία. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μπορώ να είμαι λακωνική. Να τα πω με δυο λόγια. Το παν είναι οι πολίτες. Το παν είναι οι πολίτες να μπουν στο κέντρο, στο επίκεντρο της ατζέντα μας. Το ίδιο σε ό,τι αφορά και την ανακοίνωση. Δούλεψα ως επαγγελματίας δημοσιογράφος επί δεκαετίες. Γνωρίζω λοιπόν, όσο καλός δημοσιογράφος και αν είσαι, αν η ιστορία που θες να πεις δεν είναι ενδιαφέρουσα, είναι ανώφελη προσπάθεια. Ποιος δημιουργεί τις ιστορίες, η πολιτική. Επομένως, καταρχά πρέπει να μπορούμε να πούμε ενδιαφέρουσε ιστορίες. Δεν μπορεί κανείς έπειτα να πει μια ιστορία εν κενό. Γιατί είναι ψυχρή ιστορία. Ε, δεν θα ενδιαφέρει τους ανθρώπους. Θα πρέπει να τις συνδέσουμε, τις ιστορίες αυτούς, με ανθρώπους, με πρόσωπα. Και αυτοί που λένε τις ιστορίες, οι πολιτικοί δηλαδή, εσείς δηλαδή, όταν λέτε ιστορίες τους ψηφοφόρους σας, στην εκλογική σας περιφέρεια ή εγώ, όταν πάω να πω το παραμύθι που φτιάξαμε στην Κομισιόν, θα πρέπει να συνδέσω την ιστορία με ένα πρόσωπο, με, μια προσωπικότητα, για να καταλάβει ο κόσμος ε, γιατί γράφτηκε αυτή η ιστορία. Έπειτα υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. ότι αν υπάρχουν πολλές ιστορίες που πρέπει να υποθούν, είναι σαν να μιλές καμία. Αν συνέχεια λέμε ιστοριούλες από εδώ, παραμυθάκια από εκεί, ο κόσμος τελικά βουλιάζει από το πλήθος των ιστοριών και το μόνο που θα απομείνει στο μυαλό του είναι μία οχλοβοή, αλλά όχι δεν θα κρατήσει την ουσία κανείς. Τώρα, η ανακοίνωση για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει ένα πλαίσιο τεχνικό. Στις 4 Νοεμβρίου του 2010 σας έγραψε για αυτή την ανακοίνωση εδώ στο Κοινοβούλιο. Λάβατε αυτή την επιστολή και νομίζω την έχετε στου φακέλους σας. Εκεί ανέφερα τους αδρούς άξονες, τις, βα... τις βασικές ιδέες. Δεν μιλάω για στρατηγική τώρα, δεν μιλάω για πολιτική. Μιλάω για βασικά εργαλεία. Η, Κομισιόν είναι εργα... η, συγγνώμη, η ανακοίνωση είναι, μια ένα εργαλείο ούτω ώστε να περάσει και να γίνει κατανοητό το μήνυμα. Τώρα, τούτου λεχθέντος, μπροστά στα έδρανά σας έχετε την επιστολή της 4ης Νοεμβρίου του 2010 Έχετε επίση ένα κείμενο για τους εθελοντές και έχετε και ένα έγγραφο για τους πολίτες. Έχετε δηλαδή ένα χείρας τα θέματα για τα οποία θα μιλήσω. Το 2011 θα γνωρίζετε ότι η Κομισιόν θα εστιάσει στις πολιτικές προτεραιότητες η Προεδρία έχει έρθει και σας έχει μιλήσει. Έχει εκφωνήσει την επίσημη ομιλία για της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τις βασικές προτεραιότητες τα επόμενα χρόνια. Μερικές από αυτές τις προτεραιότητες είναι βραχυπρόθεσμας. Κανένας δεν πίστευε ότι η κρίση θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της ε, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε για την κρίση βραχυπρόθεσμα. Επομένω, ανάπτυξη και θέση απασχόλησης, πολύ σημαντικά θέματα, αλλά και οι πολίτε. Οι πολίτε θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο μέχρι τις νέες εκλογές. Ξεκινάμε φέτος με, το... με ένα θέμα που αφορά την ηθαγένεια. Μιλάμε για τους εθελοντές. Εκατό εκατομμύρια εθελοντές από όλη την Ευρώπη. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι είναι εθελοντές, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί νέοι εθελοντές, νεαροί. Θα πρέπει λοιπόν φέτος ο κόσμος να αρχίσει να ενθουσιάζεται, να θέλει να ακολουθήσει να συνταχθεί μαζί μας προς την κατεύθυνση που σκιαγραφούμε. Και για να περάσουμε αυτό το μήνυμα θα πρέπει όχι μόνο να επικοινωνούμε από τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να πάμε επί τόπου και να μιλήσουμε με τον κόσμο, τον απλό κόσμο. Και μάλιστα να μιλήσουμε με διαφορετικό τρόπο στο Λουξεμβούργο και διαφορετικό την Νότια Ισπανία. Πρέπει να προσαρμοστούμε και πρέπει να προσαρμόσουμε την ιστορία μας, την ίδια ιστορία, στα αισθήματα ε, των ανθρώπων, ε, στις αντιλήψεις τους, στον πολιτισμό τους ε, και σε αυτή την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ανακοίνωση που θα ανακοινώνουμε από πάνω. Το μήνυμα αυτό, οι βασικές ιδέες υπάρχουν βέβαια και είναι οι ίδιες, αλλά το μήνυμα θα πρέπει να δοθεί επί τόπου. Και θα πρέπει να εμπλέξουμε και τις εθνικές, ε, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Και γι' αυτό έχουμε και διάφορες πλατφόρμες για να έρθουμε σε επαφή ε, με τις ε, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Ξέρετε για τους δημόσιους χώρους, ξέρετε για τα κέντρα ενημέρωσης στην Ευρώπη. Ξέρετε για τις εταιρικές ε, σχέσεις, τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που υπάρχουν σε 21 κράτη-μέλη και που με τρόπο ε, φέρνουν κοντά τους ανθρώπους που τοπικά είναι υπεύθυνοι για την ανακοίνωση. Έχουμε 13 εκπροσωπήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέονται με τα γραφεία ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία από αυτό. Εμπλέκουμε και τους βουλευτές έτσι, που είναι τα πρόσωπα. Μαζί με τους επιτρόπους της κάθε χώρας, στο εν λόγω, στο κάθε κράτος μέλους, και πηγαίνουν στις διάφορες περιφέρειες για να διαμηνήσουν όσα θέλουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα γίνει ακόμα πιο σημαντικό το, για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Στο φάκελό σας έχετε τις πληροφορίες για τις εκστρατείες αυτές εθελοντισμού οι οποίες ε, και πότε θα λάβουν χώρα στο δικό σας κράτος μέλος. Εποφεληθείτε και μεταβείτε εκεί, έρθετε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, με τους υποψήφιους εθελοντές, γιατί φέτος θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό το νήμα, να ξετυλίγεται και τα επόμενα χρόνια θα είναι τα χρόνια της ε, ενεργούς γύρανσης. Έχετε ήδη ξεκινήσει να συζητάτε το θέμα αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πάει στην Ολομέλεια του Απριλίου. Δεν θα αποφασίσουμε μόνο πόσα χρήματα θα δοθούν σε αυτά τα προβλήματα των ενεργών γυρατιών, αλλά και στις κοινωνικές πτυχές των πολιτών. Και θα παρουσιαστούν όλα αυτά το 2012. Το 2013 αν συμφωνείτε, θα είναι το έτος των πολιτών. Και γιατί. Πέρυσι προετοίμασα την έκθεση για τους πολίτες. Με όλα τα στοιχεία, τα απτά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να επιλύσουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να επιλύσουμε τα προβλήματα και ούτω ώστε οι πολίτε μα, είτε είναι τουρίστε, είτε είναι φοιτητέ, είτε θέλουν να εργαστούν σε μια γειτονική χώρα, να μπορούν να το κάνουν με πιο εύκολο τρόπο. Έχω προτείνει διάφορες νομοθετικές δράσεις, ούτως ώστε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις. Η αντίληψη θα πρέπει να είναι ότι εγώ έχω τα ίδια δικαιώματα στο γειτονικό κράτος μέλος με αυτά που έχω στο δικό μου κράτος μέλος. Και δεν θα πρέπει να υποστώ διακρίσεις, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσω δυσκολίες μόνο και μόνο γιατί πάω στη γειτονική χώρα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Ξέρουμε ότι στις διασυνοριακές περιοχές είναι πολύ δύσκολο να διέλθει κανείς στα σύνορα. Είναι πολύ δύσκολο οι επιχειρήσεις αυτές να περάσουν τα σύνορα. Φέτος λοιπόν έχουμε ξεκινήσει την κατάρριψη των φραγμών. Ένα προς ένα. Και θα συνεχίσουμε, ούτως ώστε το 2013 να μπορείτε να πείτε αυτές τις ενδιαφέρουσες ιστορίες, που είναι η χρονιά πριν τις εκλογές. Όλοι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και να πάμε να εξηγήσουμε στους πολίτες στην περιφέρειά μας, στην περιοχή μας, την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Επομένως, το Μάρτιο θα παρουσιάσω το πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Έτος για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πριν το καλοκαίρι θα έχετε το κείμενο επιτάπητος και θα ήθελα μαζί σας να ετοιμάσουμε όχι μόνο τη χρονιά αυτή το έτος δηλαδή για τους πολίτες το 2013, αλλά να έχουμε και να, κινητοποιήσουμε, και να κινητοποιηθούμε με προπαρασκευαστικές δράσεις για να είμαστε έτοιμοι το 2013. Η συνεισφορά σας ως ευρωβουλευτές που γνωρίζετε τους πολίτες, που είστε σε επαφή με αυτούς, με τους ε, εκλογεί σα, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα μας βοηθήσει τα μάλλα. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, να δούμε και την έκθεση πολιτότητας την οποία έθεσα στις 27 Οκτωβρίου και εκεί περιλαμβάνονται όλα. Όλο το πρόγραμμα εργασίας, όλος ο κατάλογος των εργασιών που πρέπει να γίνουν για να εξαλειφθούν τα, οι φραγμοί. Οι περισσότεροι φραγμοί ε, δεν είναι θεαματικά πράγματα. Είναι, για παράδειγμα, η ελεύθερη διακίνηση των εγγράφων, των πιστοποιητικών γεννήσεως, πιστοποιητικών γάμου, τέτοια ζητήματα. Επίσης, στον τομέα της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχω ήδη προτείνει και που ήδη έχει προταθεί στο Κοινοβούλιο, η εξάλληψη του εξεκουάτου ε, δηλαδή οι δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε μια χώρα να μπορούν να μεταδίδονται χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς υψηλό κόστος σε γειτονική χώρα. Τόσα πολλά στοιχεία όπως και αυτό, στοιχεία τα οποία μπορούμε μπορείτε εσείς να εξηγήσετε στους πολίτες σας, γιατί είναι χειροπιαστά, ε, αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Όταν αναλύω τι γνωρίζουν οι πολίτες για την Ευρώπη και τα δικαιώματά τους, διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλά κενά στις γνώσεις αυτές, στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Και αν δεν γνωρίζεις ποια είναι τα δικαιώματά σου, δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Γι' αυτό είναι απόλυτα σημαντικό όχι μόνο να εξαλείψουμε τα εμπόδια και τους φραγμούς, αλλά να ενημερώσουμε το κοινό ότι τα έχουμε εξαλείψει, έτσι ώστε να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Και η έρευνα που πραγματοποιήσαμε δείχνει ότι λιγότερο από ένα τρίτο θεωρούν ότι είναι καλά ή πολύ καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό μπορεί να το δείτε ως σκάνδαλο. Εγώ το βλέπω ως ευκαιρία. Σημαίνει ότι μπορούμε να κτίσουμε σε αυτό το 1 τρίτο και να ενημερώσουμε καλύτερα τα άλλα δύο τρίτα από τώρα, διότι έχουμε το χρονικό ε, περιθώριο να κάνουμε καλύτερα αυτή τη δουλειά και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό δεν αφορά μόνο λίγους πολίτες. Υπάρχουν σχεδόν 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ζουν σε διαφορετικό κράτος μέλος από το κράτος μέλος ε, καταγωγής τους και το 54% λένε ότι θα θέλανε πολύ να δουλέψουν ή να κατοικήσουν σε ένα κράτος μέλος αλλά φοβούνται γιατί δεν είναι βέβαιοι ποια είναι τα δικαιώματα τους. Γι' αυτό ε, δεν το κάνουν τελικά. Ε, δεν θέλουμε βέβαια να οθήσουμε ε, τον κόσμο να μετακομίσει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, δεν είναι αυτό που έχουμε κατά νου. Αλλά θέλουμε να τους δώσουμε την, ευκαι... την ελευθερία και την ασφάλεια εάν έχουν τέτοια πρόθεση ή αν το έχουν κάνει, αν έχουν μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος, να μην υποστούν διακρίσεις ξανά και να τύχουν σεβασμού ως Ευρωπαίοι πολίτες όπου και να βρίσκονται. Τώρα, πώς θα ενημερώσουμε καλύτερα τους ε, πολίτες, εκτός από τον άμεσο τρόπο ε, τον οποίο ακολουθείτε εσείς κάθε φορά στις εκλογικές σας περιφέρειες. Έχουμε το, το Europe Web Portal με πολύ πρακτικές πληροφορίες και σαφείς πληροφορίες και θέλω αυτό να είναι ένας σταθμός, δηλαδή εσείς ως πολίτης πάτε σε αυτό το πόρταλ και από εκεί ε, σας καθοδηγούν σε άλλα, άλλες θύρες για να απαντηθούν τα ερωτήματά σας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς οργανώσαμε αυτό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πόρταλ. Ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει ότι πάω, υποβάλλω το ερώτημά μου και θα βρω απάντηση η ελεύθερη γραμμή Europe Direct, όπου υπάρχουν ε, τηλεφωνητές που απαντάνε σε οποιαδήποτε γλώσσα Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα καλό σύστημα, λειτουργεί καλά, θα προσπαθήσω να το απλουστεύσουμε. Όλα ξεκινάνε με έναν αριθμό τηλεφώνου, είναι ένας μεγάλος αριθμός που δεν τον θυμάται ε, κανείς, είναι, είναι σημαντικό, δεν είναι απαραίτητο είναι ε, πιο σημαντικό να πάρεις την απάντηση όταν τηλεφωνήσεις, αλλά θα πρέπει να απλουστεύσουμε τον τρόπο πρόσβασης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης ε, τα 500 κέντρα, τα τοπικά κέντρα πληροφόρησης για την Ευρώπη επίσης κάνουν καλά τη δουλειά τους. Όλα αυτά θα πρέπει να ε, συνδεθούν έτσι ώστε το 2013 να έχουμε φτιάξει ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο που να μας βοηθήσει να μεταδώσουμε τα μήνυματα και να μας ε, βοηθήσει να βοηθήσουμε τους πολίτες να ε, λάβουν τα μηνύματα που ζητούν. Όταν ανακοινωθούν οι δράσεις ε, σε αυτή την έκδοση θα, ε, θα, θα αξιολογήσουμε την πρόοδο, θα ε, καταρτήσουμε ένα σχέδιο δράσης για να εξαλείψουμε όλα τα αναπομείναντα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν ασκούν τα δικαιώματά τους. Πρόεδρε, λοιπόν, μέχρι στιγμής κανείς ε, εδώ στο Κοινοβούλιο, καμία επιτροπή του Κοινοβουλίου δεν έλαβε, ε, δεν ανέλαβε αυτή την έκθεση για τον πολίτη. Είναι μια ε, γκάρσια ε, έκθεση γιατί αφορά τα πάντα στη ζωή. Είναι μια έκθεση για την εσωτερική αγορά. Είναι μια έκθεση για την πολιτισμική διαφορετικότητα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τα πάντα όσα αφορούν τον πολίτη, τη ζωή του πολίτη ε, θα, πρέπει κανείς να ε, προετοιμάσει μέσα από αυτή την έκθεση το έτος για τον πολίτη που θα παρουσιάσω σε μια πρόταση που θα εκδοθεί φέτος τον Μάρτιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρέντινγκ. Τώρα έχουμε κάποιους που θέλουν να διατυπώσουν κάποιες ερωτήσεις. Ο Πεγκάντ, κυρία Βεζέ, τον κύριο Κορέα, Κορία, Φαρσάκε και συνεχίστε, σημειώνετε τα ονόματα. Λοιπόν, όλοι θα λάβετε τον λόγο. Βαργάρτ, παρακαλώ. Thank you, and I will do this in uh, Danish. Θα μιλήσω δανέζικα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, στο κανάλι 6 για να μ' ακούσετε. Σας ευχαριστώ που μας επισκεφτήκατε στο ταπεινό μας κοινοβούλιο. Είναι πολύ ευχάριστο που ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για την πολύ συγκεκριμένη και πολύ εστιασμένη παρουσίασή σας για τα προγράμματά σας, για τα σχέδιά σας τα επόμενα χρόνια. Σέβομαι πάρα πολύ το ρεαλιστικό σας πνεύμα, το πρακτικό σας πνεύμα. Ε, άκουσα στην παρουσίασή σας με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Και εγώ ήμουν δημοσιογράφος επί δεκαετίες. Ίσως γι' αυτό λοιπόν να συμφωνούμε τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση, ίσως και εσείς να την έχετε, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που λείπουν. Είναι ένας τεράστιος τομέας αυτός. Δεν είναι κάτι που ένας μόνο επίτροπος ή μία επιτροπή μπορεί να καταφέρει. Πρέπει να συνεργαστούμε για να υλοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους. Το Σεπτέμβριο για αυτή την έκθεση προσπάθησα να με... Συγκεκριμένο όταν πήρα το λόγο. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στην επιστολή της 4ης Νοεμβρίου. Νομίζω ότι είναι σωστό ότι δεν πρόκειται για στρατηγική. Αυτό το κείμενο, αυτή η ανακοίνωση δεν είναι μια απλή στρατηγική. Συμφωνώ. Πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό από μια στρατηγική. Α την ονομάσουμε σχέδιο δράση. Όπω θέλετε, επίτετη. Το έγγραφο αυτό, και δεν ξέρω πόσοι το διάβασαν, εγώ πάντως το διάβασα, είναι ένα πολύτιμο έγγραφο εργασίας. Με πολλά καλά στοιχεία. Είναι ουσιαστικά μια περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε. Είναι μια περιγραφή των στοιχείων τον οποίο, τα οποία έχουμε ήδη δρομολογήσει. Και τώρα πάω στην ερώτησή μου. Και θα προσπαθήσω να τη διατυπώσω τόσο συγκεκριμένα όσο ήσασταν και εσείς στην παρουσίασή σας. Ας ονομάσουμε λοιπόν αυτό το κείμενο σχέδιο δράσης. Ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει ένα όραμα για το πού πάμε, χάρη στην ε, συλλογική δουλειά της ε, Επιτροπής, υπάρχει μια συμφωνία του 2008 που συμφωνήσαμε να κινηθούμε προς την ίδια κατεύθυνση για τον κοινό μας στόχο. Θα ήθελα να υπάρξουν δύο λόγια για το όραμά μας. Συμφωνώ με τους στόχους και τις φιλοδοξίες και τις επιθυμίες πολλών ε, συναδέλφων στο Κοινοβούλιο. Αλλά θα ήθελα ένα όραμα. Και επίσης αυτό το διευρυμένο έγγραφο να μιλήσουμε για τα κοινωνικά ΜΜΕ που χρειαζόμαστε στο πλευρό μας για να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα όραμα λοιπόν, το οποίο αγκαλιάζει όλα τα θέματα και εστιάζει στον κοινωνικό ρόλο των ΜΜΕ. Μπορεί η Κομισιόν να το συμπεριλάβει αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Σας ευχαριστώ κύριος παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι ας το πούμε έτσι τα δικαιώματα των πολιτών, όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, έτσι, έτσι το αποκαλούμε. Μετά όμως έχουμε μετά το όνομα, έχουμε και το επώνυμο. Είμαι Ευρωπαίος πολίτης, είμαι καλλιτέχνης, είμαι φοιτητής, είμαι καθηγητής, δικηγόρος, ε, είμαι ο αυτοκινητιστής. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εδώ αρκετές, πολλές, ε, πολλοί περιορισμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή για πολλά επαγγέλματα που θέλουμε να ασκήσουμε παντού στην Ευρώπη. Σήμερα το πρωί είχαμε του υπουργού από την Ουγγαρία, την Ουγγρική Προεδρία και θίξαμε το θέμα τη κινητικότητα των καλλιτεχνών στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, σε κάποιες χώρες πρέπει να έχουν θεωρήσει διαβατηρίων. Τι γίνεται με την κοινωνική του ασφάλιση, για παράδειγμα. ένα μουσικό που παίζει στην ορχήστρα μια χώρα, όταν πάει σε ορχήστρα άλλη χώρα, τι συμβαίνει με όλα αυτά. Είναι θέματα λοιπόν που ακόμα υπάρχουν πολλοί περιορισμοί, όροι και προποθέσει Ίσως ε, ακόμα και μπορώ να θυμηθώ το ότι όταν ήμουν στη Σλοβενία ζητούσαν ένα αυτοκόλλητο σήμα για τα αυτοκίνητα για να μην ε, υποστούν ε, ένα πρόστιμο. Σε άλλες χώρες δεν ζητείτε κάτι τέτοιο. Δημιουργείται έτσι μια σύγχυση σε πολλά θέματα και που δεν είναι, ας το πω, γενικά θέματα ε, τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, αλλά είναι εξειδικευμένα ξεχωριστά θέματα που αφορούν και πλήττουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και μετά ένα άλλο θέμα, το θέμα των ιδρυμάτων από ό,τι άκουσα, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που επιτρέπει να υπάρχει ένα ε, ίδρυμα που ε, μπορεί να λειτουργεί για όλες τις άλλες χώρες είναι η Ολλανδία. Για όλες τις άλλες χώρες, για παράδειγμα, ένα ίδρυμα στην Ισπανία και θέλω να εργαστώ για αυτό το ίδρυμα στο Λουξεμβούργο. Πρέπει να ζητήσω, να έχω αίτηση προς την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου που θα διατυπωθεί, να δημιουργηθεί ένα νέο τέτοιο χορηγικό όργανο, ένα τέτοιο ίδρυμα στην Γερμανία, αλλού και στις άλλες χώρες. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα για τα ιδρύματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να μπορούν ως μεκίνες, ε, ως χορηγοί να μπορούν να δράσουν. Ευχαριστώ. Κύριος Μάρκος Κορέα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο και τις εύχομαι και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους καλή χρονιά ε, και καλή τύχη στην ε, χρονιά του εθελοντισμού, την προσπάθεια που έχουμε ήδη ξεκινήσει και για την οποία μας μίλησε. Καλή τύχη και σε όλες τις πρωτοβουλίες που μας ανέφερε. Θα ήθελα να πω ότι μου αρέσει όλος ιδιαίτερος η λεπτομέρεια με την οποία ε, προωθεί η Κομισιόν και στα 27 κράτη-μέλη για να ακούσει ιδέες και από τα 27 κράτη-μέλη και να προωθήσει τις ιδέες της. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε η Επίτροπος, να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες, να έχουμε μία σχέση με τις επιχειρήσεις, με τις τοπικές οργανώσεις κτλ. Για αυτή την, ε, αυτό το κείμενο της ανακοίνωσης, κύριε Ρέντινγκ, ακυρώθηκε ένα πρόγραμμα, ε, η χρηματοδότηση μάλλον ενός προγράμματος για την ε, λειτουργία ενός ε, ευρωπαϊκού καναλιού. Σε αυτό το τομέα υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προσπαθήσει, είχαν αρχίσει να δουλεύουν για να στηθεί αυτό το κανάλι. Η Ευρώπη υποτίθεται ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους πολίτες. Τι εναλλακτική λύση έχει η Κομισιόν, μια και ακυρώθηκε αυτή η χρηματοδότηση και μια και δεν προχωράει, δεν θα προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα. Η κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Για, το θέμα, για μένα το θέμα της ηθαγένειας είναι θεμελιώδες. Είναι ένα θέμα οριζόντιο και καθολικό Εξού και η δυσκολία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί πραγματικά και να εναγκαλίσει αυτή την, αυτό το ζήτημα. Είναι όμως σημαντικό αν θέλουμε οι πολίτες να ενδιαφερθούν επιτέλους για τα ευρωπαϊκά διακυβευόμενα. Ε, μ' άρεσε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πολλές πληροφορίες είναι σαν να μην δίνουμε καμία πληροφορία τελικά, ισοδυναμεί με αυτό. Ε, ισχύει αυτό. Όταν εγώ συζητάω με τους Ευρωπαίους πολίτες ε, σε διάφορες συζητήσεις, μας λένε το εξής, μας λένε ότι οι πληροφορίες είναι απροσπέλαστες, δεν ξέρουν πού να τις ψάξουν, υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες που μπορεί κανείς να, να ενημερωθεί, ας πούμε, που τελικά η πληροφορία δεν περνάει, που τελικά δεν ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί μπορεί να ψάχνει από εδώ, από εκεί, από και παρακεί. Τελικά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έχουν χάσει τον μπούσουλα, τον μπούσουλα και πιστεύουν ότι οι αποφάσει των Βρυξελών του πέφτουν στο κεφάλι. Ε, το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σα πω Νομίζω ότι θα πρέπει να βγούμε από αυτό το ευρωπαϊκό μας γυάλινο πύργο. Έχω υπόψη μου τι συζητήσεις που οργανώνουν αυτά τα ενημερωτικά κέντρα, τα κέντρα πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα γραφεία, αν θέλετε καλύτερα, ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα γραφεία αυτά τα οποία εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτά δυσκολεύονται να οργανώσουν ε, συζητήσεις και να ενδιαφερθούν κι άλλοι πέρα από αυτού που ούτω ή άλλω ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά θέματα. Το θέμα είναι πώ θα κινητοποιήσουμε του πολίτε. Πώ ε, θα φτάσουμε πιο κοντά σε αυτού. Ο κ. Κούρια μίλησε για την τηλεόραση, για τηλεοπτικά κανάλια. Εγώ μιλάω για τα τοπικά ραδιόφωνα, να έρθουμε σε επαφή περισσότερο με, τα τοπικά, με την τοπική ραδιοφωνία. Κάτι άλλο που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Σκούρια. Σκούρια. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ΜΜΕ ε, με συμμετοχικό τρόπο λειτουργίας που δουλεύει με τους πολίτες και που ε, ε, ζήτησαν χρηματοδότηση από την Κομισιόν, τους, τους την αρνηθήκαμε. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Γιατί όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά τα ζητήματα δεν ανταποκρίνονται σε καμία γραμμή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δηλαδή, τα περνάμε από τη μία γραμμή του ενός προγράμματος στην άλλη γραμμή. Και τελικά αντιμετωπίζουν διαδοχικέ αρνήσει. Δεν του δίνουμε, α πούμε, δεν τα προωθούμε, δεν του δίνουμε χρηματοδότηση κτλ. Τρίτο θέμα. Διακόπτε όμω από την πρόεδρο. Α, όχι. Μου έκανε εντύπωση μία φράση. Δεν θυμάμαι σε ποιο έγγραφο την βρήκα, αλλά αναφερόταν ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι Ευρωπαίοι την ευρωπαϊκή του ηθαγένεια. Όσο βλέπουμε αυτά τα θέματα με αυτόν τον τρόπο, θα τα βλέπουμε ανάποδα. Επίσης μου κάνει εντύπωση, όταν εξηγούμε τα πράγματα στους Ευρωπαίους, μου κάνει εντύπωση το πώς πραγματικά εγείρεται το ενδιαφέρον τους. Έχουν την εντύπωση, λοιπόν, ότι οι Βρυξέλλες ή οι τεχνοκράτες των Βρυξελών λαμβάνουν τις αποφάσεις χωρίς καμία σχέση, ε, χωρίς να τους λάβουν υπόψη, χωρίς να τους δώσουν καμία πληροφορία εκ των προτέρων. Και τελικά, με αυτόν τον τρόπο, επειδή έχουμε αυτή την αντίληψη, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποια χρησιμότητα. Νομίζω επ' αυτών των θεμάτων θα πρέπει να δουλέψουμε. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε μια ηθαγένεια, η οποία να μην ξεκινάει από πάνω προ τα κάτω, αλλά να ε, δώσει. Α, να αποκτήσουν επίγνωση δηλαδή οι πολίτε για τα δικαιώματά του, ναι, μεν, αλλά να του δώσει και τη δυνατότητα να εκφραστούν, από κάτω προ τα πάνω δηλαδή. Ελπίζω να μην ξεγελάσουμε τους πολίτες Ελπίζω να... ότι είναι σημαντικό αυτό για να ανέβει η συζήτηση από τη, βάση προς τα πάνω. Κάτι άλλο. Καλό του συναδέλφου μου να υπογράψουν την δήλωση 84, υπαριθμών 84, που ζητάει ε, να υπάρξει συγκεκριμένο καθεστώς για όλα τα, αυτά τα ιδρύματα και για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα να υπάρξει ένα νομικό καθεστώ σαφέ. Ένα θα παρέμβει ακόμα και μετά μπορεί να αρχίσει με τι απαντήσει η κυρία Ρέντινγκ. Ο συνάδελφο Ιβαν, παρακαλώ. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή στη διαφορά που υπάρχει και αυτό το γνωρίζω και από τη δική μου εμπειρία ανάμεσα στην σωστή επικοινωνία και αποτελεσματική επικοινωνία μπορούμε να γράψουμε ολόκληρε διατριβέ για το πώ μπορούμε να επικοινωνούμε. Σίγουρα θα βρούμε εμπειρογνώμονε σε επίπεδα επιτροπής, κρατών μελών για το πώ θα πρέπει να επικοινωνούμε σωστά και να μεταδίδουμε σωστά τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι αυτές οι διατριβές και τα δοκίμια θα είναι πάρα πολύ βαρετά και ανιαρά τελικά ενώ μια αποτελεσματική ανακοίνωση, η ενημέρωση είναι μια δημιουργική πάνω απ' όλα γιατί οι πολιτικές αυτά που κάνουμε εδώ για να υποστηριχθούν από τους πολίτες της Ευρώπης θα πρέπει αυτό που κάνουμε εμείς εδώ να είναι ενδιαφέρον για τους πολίτες. Πέρθη είχαμε 50 δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, δημοσιογράφους από τη Ρουμανία που ε, μπλέκονταν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και πήγαμε με τον Σαντιαγκο Φίσας, με τον Λόκεγκαρτ και με την Πέτρα Κάμερβερτ και συζητήσαμε αρκετές ώρες μαζί τους και στο τέλος μας είπαν πολύ, με μεγάλη ειλικρίνεια και αμεσότητα ότι αν είχαν να γράψουν ένα άρθρο για αυτή τη συζήτηση δεν θα μπορούσαν να γράψουν κάτι. Είναι σαφές ότι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι για αυτούς που γνωρίζουν πολύ ενδιαφέρον. Οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είναι ειδικοί στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η πλειοψηφία δεν γνωρίζουν ποια είναι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς λειτουργούν όλο το σύστημα, το, τις διαδικασίες. Δεν ε, διακρίνουν ανάμεσα στην εθνική κυβέρνηση και το Εθνικό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα, αν εμείς θέλουμε να μας υποστηρίξουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί χρειαζόμαστε αυτή την υποστήριξη, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Πρέπει να δείξουμε κάποιο ενδιαφέρον. Γιατί ένα άρθρο στον τύπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση το διαβάζει κανείς μόνο αν έχει ενδιαφέρον. Ε, πάει κανείς στη βιβλιοθήκη και ψάχνει κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν τους ενδιαφέρει αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό θα πετύχουμε να είμαστε και δημιουργικοί, όχι μόνο σωστοί στη μετάδοση των μηνυμάτων και να κάνουμε τη δραστηριότητά μας πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα η κυρία Σάκα, είχε ζητήσει τον λόγο στην αρχή. Στον επόμενο γύρο, εντάξει, γίνεται. Λοιπόν, έχετε τον λόγο κυρία Ρέντινγκ. Όχι, εσείς ε, ευχαριστώ πολύ και που ζητήθηκε η παρέμβαση. Λοιπόν, κατανοώ θα έλεγα αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες και υπάρχει μια συμφωνία που είναι αρκετά γενικευμένη μεταξύ αυτών που παρενέβησαν και τις Επιτροπής και δεν πρόκειται εδώ για μεγάλα θεσμικά ή θεωρητικά ζητήματα και για τους δημοσιογράφους εκτός αυτών που βρίσκονται εδώ στις Βρυξέλλες και που δεν θα κατανοούσαν τίποτα για όλα αυτά και ούτε συνδέεται άμεσα στη ζωή με τη ζωή των πολιτών. Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος ακριβώς για τον οποίο υπέβαλα στην εισαγωγική μου παρουσίαση τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι πρέπει να έχουμε τα πολύ συγκεκριμένα χειροπιαστά στοιχεία για να επεξηγήσουμε στους πολίτες μας τι κάνει ακριβώς η Ευρώπη στο ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτούς. Δίνω αυτό το παράδειγμα, όχι επειδή το έκανα εγώ ίδια αυτό, αλλά επειδή όλοι σας ε, είχατε πάει στις ευρωεκλογές ε, και ε, γνωρίζετε το τι συνέβη σε σχέση με την τελευταία περίοδο. Ήταν κάτι λοιπόν το οποίο κατανοούσαν οι πολίτες, το κατανόησαν με σαφήνεια, διότι τους αφορούσε άμεσα στην καθημερινή τους καθημερινή ζωή. Ακριβώς αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και να συνθέσουμε και να πετύχουμε στην δράση για τους πολίτες. Αυτό που κάνει η Ευρώπη στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που δεν μπορεί να γίνει σε ένα επίπεδο κρατών μελών, σε εθνικό επίπεδο, για να επιληθούν τα διασυνοριακά θέματα μεταξύ των κρατών σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να είναι ένα θέμα να θέλει κάποιο να πάρει το αυτοκίνητό του όταν όταν πάει σε μια γειτονική χώρα τι κάνει κανείς, να παίρνει κανείς ε, δύο φορές ε, ταξί και να χρησιμοποιεί όλη τη γραφειοκρατική επιβάρυνση που υφίσταται, γιατί μην το κάνουμε πιο απλά και εύκολα. Το κάναμε αυτό. Σε σχέση λοιπόν ε, με τον τρόπο αυτό δείχνουμε, κοιτάξτε πολίτες, με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ζωή σας πιο απλή και πιο αποτελεσματική. Ή για παράδειγμα ένας τουρίστας που έχει εμπλακεί σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα, σε ένα ατύχημα σε μια γειτονική χώρα. Τον, πιάνει, τον παίρνει η αστυνομία, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει τα θέματα των δικαιωμάτων των ατόμων που συλλαμβάνονται από την αστυνομία και οδηγούνται στα κρατητήρια, στις φυλακές. Θα υπάρχει μια δέσμη ελάχιστων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη που αυτόματα θα ισχύουν ως δικαιώματα για τους πολίτες. Αυτόματα θα μπορούν να πληροφορηθούν τι τους συμβαίνει, ποια είναι η κατηγορία που τους εγείρεται, που διατυπώνεται εις βάρος τους και μάλιστα όλα αυτά στη γλώσσα τους. Και όλα αυτά βρίσκονται υπό εξέλιξη, ενρευστό, εξελίσσονται και αναπτύσσονται. Πολλά παραδείγματα θα μπορούσα να σας αναφέρω συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, έχετε αυτό τώρα στο φάκελό σας, αυτό το fish, τι σημαίνει αυτό. Κάποιες νομικές αποφάσεις αυτές, σε αυτά τα δελτία FISH, δελτία όσον αφορά προτάσεις που βρίσκονται καθοδόν και θα έχουν διευθετηθεί ε, στο, θα διευθετηθούν στο μέλλον. Μέχρι το 2013 λοιπόν πολλά από αυτά τα πράγματα, τα προβλήματα, τα συγκεκριμένα και χειροπιαστά και που συσχετίζονται με την καθημερινή ζωή των πολιτών θα έχουν επιληθεί, θα έχουν διευθετηθεί. Σας δίνω ένα παράδειγμα για το τι έγινε σε σχέση με τον τελευταίο μήνα. Ένα από τα στοιχεία τα οποία είχαν περισσότερο αναφερθεί στο εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο από δημοσιογράφους στον τύπο ήταν το θέμα των διαζυγίων όσον αφορά μεικτούς γάμους ή διεθνείς εντός εισαγωγικών γάμους. Κάποιος Γάλλος έχει παντρευτεί στην Πολωνία, ζουν, μια Πολωνέζα ζουν στο Βέλγιο, για παράδειγμα, διαλύεται ο γάμος, διαζύγιο, τι γίνεται στη συνέχεια. Πολύ συγκεκριμένα. Πώς επιλύουμε το πρόβλημα, όχι το πρόβλημα, αλλά τι κάνουμε με το διαζύγιο, πώς ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα αν υπάρχει απόφαση να έχει ληφθεί απόφαση να πλουστευτεί η ζωή τους τι γίνεται με πιστοποιητικά γέννησης κτλ. Κοιτάξτε αυτά τα δελτία fish κοιτάξτε την έκθεση για τους πολίτες θα δείτε ότι δίνονται απαντήσεις δεν επαρκούν όλα αυτά βέβαια όπως είπα και στην εισαγωγή μου να κάνουμε μόνο αυτά Πρέπει επίσης να κάνουμε τους πολίτες να αντιληφθούν ότι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, ότι έχουν όλα αυτά τα νέα δικαιώματα. Και γιατί έχουν όλα αυτά τα νέα δικαιώματα. Επειδή διότι υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο αποφάσισε να υφίστανται αυτά τα δικαιώματα και να μπορούν να τα διεκδικούν. Αυτό επιθυμούμε ακριβώ. Εκείνοι οι οποίοι πάνε στι ευρωεκλογέ το 2014, 14 δεν είναι νομίζω, να μπορούν να μιλήσουν, να πούνε στους πολίτες, ειδού να τι κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το άλλο και το παρακάτω άλλο πρόβλημα επιλύσαμε και διευθετήσαμε, ώστε να έχετε εσείς πολίτες περισσότερα δικαιώματα. Αυτό είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους ε, για τους πολίτες. Και αυτό δίνει απαντήσεις επίσης ε, στα ερωτήματα που αντιμετωπίζονται και διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι. Διότι δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος σε αυτό το επίπεδο, στον περιφερειακό τοπικό τύπο, πρέπει να έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο στα χέρια του, που να συσχετίζεται με την καθημερινή ζωή των πολιτών. Για παράδειγμα, έδωσα αυτό το δελτίο σε σχέση με τους επιτρόπους όταν πάνε κάπου σε κάποια περιφέρεια, σε κάποια περιοχή, όχι μόνο να μιλήσουν για το θέμα το οποίο έχουν να παρουσιάσουν, αλλά να πούν, για κοιτάξτε εδώ για παράδειγμα, με αυτό με το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης, αυτό το μέσο, με αυτό το σχολείο, αυτό το δρόμο, αυτή την προσπάθεια ας πούμε διατήρησης, ε, συντήρησης της φύσης, ε, συγχρηματοδοτήθηκαν όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκονται στη γειτονιά σας. Πρέπει να πάμε στο τοπικό επίπεδο, γιατί διαφορετικά δεν θα ενδιαφερθούν οι δημοσιογράφοι με άλλο τρόπο για τέτοια θέματα. Έχω τον στόχο, για παράδειγμα, από τη στιγμή που ξεκίνησα να ε, έχω σχέση με τα θέματα της Ιθαγένειας και των πολιτών ως χαρτοφυλάκιο δικό μου, να καταφέρω να έχουμε θετική απήχηση στους τίτλους και στα δημοσιεύματα του τύπου σε εφημερίδες και τύπο που είναι δημοφιλής. Μια, ας το πω έτσι, ένας θετικός τίτλος φιλευρωπαϊκός στην Bildzeitung στη Γερμανία, μια λαϊκή εφημερίδα. Είναι δυνατόν και εφικτό να γίνει αυτό με τέτοια μικρών διαστάσεων εγχειρήματα. Μπορούμε έτσι να επεξηγήσουμε στους δημοσιογράφους και να αντιληφθούν οι πολίτες ότι αυτές είναι οι καλές ειδήσει, τα καλά μαντάτα. Αυτά πρέπει να δίνονται από τους υπεύθυνους στο πολιτικό επίπεδο των Βρυξελών προς τους πολίτες. Πρέπει να αποφασίζεται το θέμα τέτοιων δραστηριοτήτων και μετά να πηγαίνουμε να περνάμε στους πολίτες επεξηγώντας ποια ήταν η απόφαση που ελήφθη και τι γίνεται. Και αυτό είναι φυσικά τα κοινά κέντρα ε, επικοινωνίας και πληροφόρησης ε, που έχουν τεράστια σημασία. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και ετών να κάνουμε κάτι παραπάνω για, μέσω αυτών. Διότι λειτουργούν καλά και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μοιράζονται κοινέ πρωτοβουλίε. Είναι κάτι πολύ ε, ελκυστικό, θελκτικό αυτό και δίνει επίσης και τη δυνατότητα να έχουμε ένα ευδιάκριτο πρόσωπο με το οποίο θα μας ταυτίζουν και μας ταυτοποιούν οι πολίτες για τα θέματα που αποφασίζονται εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μετά νομίζω ήδη εν μέρη απάντησα κάπως ε, προς τον κύριο Λόκεγκάρντ. Με μια τέτοια ακριβώς προσέγγιση είναι θα έλεγα άχρηστο να συντάσει κανείς να χαράζει μια ευρύτερων διαστάσεων στρατηγική. Διότι μια στρατηγική μπορεί να αναφερθεί ε, σε μια πρόταση. Τώρα να φτάσουμε, να περάσουμε στους πολίτες και να επεξηγήσουμε τις αποφάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εμπλέκει αυτή την προσέγγιση. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε όχι στρατηγική, αλλά μέσα και εργαλεία που είναι αποτελεσματικά. Ένα από αυτά τα εργαλεία, και έχετε απόλυτο δίκιο φυσικά για αυτή τη δουλειά, είναι τα νέα μέσα. Τα κοινωνικά δίκτυα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν τα χρησιμοποιούμε επαρκώς όσο πρέπει προβληματιζόμαστε και θα δούμε μαζί από κοινού πώς μπορούμε να επιβάλλουμε την χρήση, την χρησιμοποίηση αυτών των νέων μέσων Ποτέ δεν θα σκεφτόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσα κάποτε να έχω εμπλακεί στο Twitter. Αλλά τα μέλη της, του γραφείου μου με εξοικείωσαν και κατάφερα και σε αυτό να προσέλθω. Χρειαζόμαστε αυτά τα νέα μέσα λοιπόν για να προσεγγίσουμε τους πολίτες. Και πρέπει να τροφοδοτήσουμε, να δώσουμε στοιχεία στους ε, δημοσιογράφους που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Τι κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναέτος χιλιάδες ε, δημοσιογράφους ε, μεριμνά για αυτούς που προσέρχονται για να καταρτιστούν και να εξηγηθούν να μάθουν για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Γίνεται με πολύ αντικειμενικό βέβαια τρόπο αυτό να τους επεξηγήσουμε πώς λειτουργούν τα γρανάζια των θεσμικών οργάνων. Έχουμε χιλιάδες δημοσιογράφους που συμμετέχουν σε αυτά τα μαθήματα και σεμινάρια κατάρτισης για την μεθοδολογία και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί δεν προσέρχονται μόνο απλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έρχονται και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της μαθητείας και εξοικείωσή τους και πάνε και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Νομίζω δεν συνεργαζόμαστε αρκετά επαρκώς όπως θα έπρεπε με την Επιτροπή Περιφερειών. Και πράγματι πιστεύω στεναρά ότι οι δήμαρχοι και ότι οι πρόεδροι των μεγαλύτερων, των μεγάλων περιφερειών έχουν τεράστια σπουδαιότητα για να συνεισφέρουν να περάσει αυτό το μήνυμα προς τους πολίτες. Αυτό λοιπόν, αυτό το κοινό εγχείρημα για να προσπαθήσουμε να επεξηγήσουμε προς τους πολίτες τι κάνουμε και πώς γίνονται όλα αυτά είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και ναι κύριε Φίσας, είναι πολυσχηδή τα πράγματα σε σχέση με τους πολίτες. Και εδώ σε σχέση με αυτή την κοινοβουλευτική σας επιτροπή από κοινού <clears throat> με τον συνάδελφό μου υπεύθυνο για τα πολιτισμικά θέματα πάλι λοιπόν θα ε, ε, δοθεί συνέχεια σε ένα πρόγραμμα που είχε, ένα σχέδιο που είχε εξεταστεί πριν από περίπου 10 χρόνια το είχαμε δει. Κινητικότητα των καλλιτεχνών. Θα μπορέσουν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν μόνο όταν τα γενικότερα θέματα κινητικότητα των πολιτών θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Παρότι έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών σήμερα, εξακολουθούν και υφίστανται πολλά προσκόμματα, πολλά εμπόδια σε αυτή την ελευθερία. Πολλά από αυτά είναι διοικητικού χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικά πάντα νομικού πλαισίου νόμων ή ε, νομοθετημάτων. Κανένας δεν ε, πίεσε τα κράτη-μέλη να άρουν αυτά τα εμπόδια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να απαριθμηθούν, να, να τα απαριθμίσουμε, να κάνουμε ένα κατάλογο όλων αυτών των ε, προσκομμάτων που παρεμποδίζουν τους καλλιτέχνες, τους δικηγόρους, τους τουρίστες, τους φοιτητές να αντιμετωπίζονται όπως θα έπρεπε σε ένα άλλο πλαίσιο πιο ελεύθερο στην κινητικότητά τους όταν περνάνε σε μια άλλη χώρα. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει. Είναι πολλά μικρά στοιχεία που συναπαρτίζουν αυτό. Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα αυτά τα μικρότερων διαστάσεων στοιχεία, αυτές τις ψηφίδες όταν τους τις παρουσιάζουμε με βιώσιμες λύσεις, όταν τους τα παρουσιάζουμε με λύσεις που μπορούν να δοθούν για να είναι αποτελεσματικότερες, για να δοθεί μια λύση. Υπάρχουν άνθρωποι που με αφοσίωση θέλουν να βοηθήσουν να γίνει κάτι, να βελτιωθούν τα πράγματα και έχουν αντιμετωπίζονται πολλά εμπόδια πάλι εκεί. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να δούμε κατά το έτος ε, των εθελοντών είναι η διασυνοριακή εθελοντική εργασία. Γιατί δεν λειτουργούν τα πράγματα εκεί. Λόγω αυτών των προσκομμάτων των ε, φραγμών και εμποδίων. Και εδώ έχουμε πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί και πρέπει να τα εγγράψουμε όλα αυτά στον κατάλογο των ενεργειών που, και πρωτοβουλειών που θα αναλάβουμε. Και για το δίκτυο τώρα των ε, τηλεοπτικών σταθμών. Έχουμε δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών, μικρών ε, ας το πω έτσι εμπλεκόμενων και ε, λειτουργούν τα πράγματα καλά εκεί. Υπάρχει πολύ, μικρός, πολύ μικρή γραφειοκρατική επιβάρυνση για να λειτουργήσουν αυτά. Με βάση αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργεί λοιπόν καλά σήμερα είχαμε και την πρόταση να υπάρξει εκ παραλίλου και ένα δίκτυο τηλεοπτικών σταθμών για τηλεοπτικές εκπομπές. Και θα έρθω στη συνέχεια και στο θέμα των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων που συνδέεται με αυτό το πλαίσιο. Το πήρα πολύ σοβαρά και το εξέτασα σε βάθος το πρόβλημα και είδαμε ότι στη δημοσιονομική κατάσταση όπως έχει σήμερα. Οι προτάσεις αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές όσον αφορά το δημοσιονομικό τους χαρακτήρα και πλαίσιο. Θεώρησα ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να επικεντρωθούμε και να διευρύνουμε, να επεκτείνουμε φυστάμενες δυνατότητες και συστήματα ως μέσα, ως εργαλεία, παρά να δημιουργήσουμε επιπρόσθετα που στο τέλος τέλος δεν θα ήταν και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Και καμιά φορά ως επίτροπος πρέπει κανείς να παίρνει αποφάσεις. Εγώ είμαι ιδιαίτερα Λουξεμβούρια, βλέπετε σε αυτό το πλαίσιο. Είμαστε προσγειωμένοι, ρεαλιστές λέμε φέρνει κάτι, δίνει κάποιες ε, λύσεις, ε, αξίζει τα χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν, value for money, money. Αυτά τα οποία είχαμε επιτραπέζεις εδώ ως προτάσεις με οδήγησαν έφνης στο συμπέρασμα ότι καλύτερο θα ήταν να σταματήσουμε αυτή την πορεία. Όσοι ήταν, ανταγωνιζόντουσαν ή συγγνώμη, συνεισέφεραν και είχαν αναπτύξει αυτές τις προτάσεις πληρώθηκαν για το έργο που είχαν κάνει δεν ήταν ότι υπήρχε μόνο ε, η επένδυση από πλευράς χρόνου και έργου υπήρχαν και οι ελπίδες που είχαν βέβαια επενδύσει αλλά οικονομικά αποζημιώθηκαν ώστε δεν υπάρχουν πλέον κάποιες διεκδικήσεις κάποιες εκκρεμότητες ε, τώρα για τις ενισχύσεις. Έχουμε πολλές, ε, πολλά αιτήματα, πολλές αιτήσει για επιχορηγήσεις και έχουμε και πολλές αιτήσει που σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες που έχουμε και ε, διέπουν αυτό το πλαίσιο πολλά πράγματα δεν υλοποιούνται όπως θα έπρεπε. Ζήτησα από την ομάδα μου να εξετάσει το πλαίσιο όλων των επιδοτήσεων που χορηγούμε. Υπάρχουν πάμπολες και πολύ συχνά είναι, ας το πω κάτι, μια ε, δράση που δεν οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα αξιόλογο. Θα πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμιστεί όλο αυτό το σύστημα κάποια μέρα, το σύστημα των ενισχύσεων. Και σας λέω και προαναγγέλω ήδη σήμερα ότι οι μισοί από εσά θα αποστείλουν επιστολές που θα συντάξουν σε μένα. Ενώ 100% θα αναφερόταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ε, η προσπάθεια να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες και να αξίζουν τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται. Θα έχουμε σίγουρα, κυρία Πρόεδρε, είμαι βέβαια μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα αυτά. Θα έχετε κατανοήσει εν τω μεταξύ ότι θα ήθελα όλα αυτά να είναι βιώσιμα και λειτουργικά. Κατά το τέλος αυτής της περίοδου να έχουμε όταν θα πρέπει να πάμε στους πολίτες να λογοδοτήσουμε να πούμε ειδού τι κάναμε να έχουμε ισχυρά επιχειρήματα ισχυρά επιχειρήματα με βάση τις δράσεις που θα έχουν ε, γίνει. Και δεν θα είναι η Επίτροπος ή ο Επίτροπος μόνο που θα το κάνει αυτό. Όλο το Κοινοβούλιο, όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές στις επόμενες ευρωεκλογές θα πρέπει με αυτά τα, αυτά τα, αυτά τα θέματα αυτού του χαρτοφυλακίου να μιλήσουν προς τους πολίτες. Ας τα κάνουμε λοιπόν από κοινού όλα αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε 11 συναδέλφους που έχουν ζητήσει να παρέμβουν και να διατυπώσουν ερωτήσει. Να μην κάνετε πολλά σχόλια γιατί διαφορετικά δεν θα τελειώσουμε. Πρέπει στι πέντε να ολοκληρώσουμε. Ερωτήσεις λοιπόν να διατυπώνετε. Η κυρία Σάκρε παρακαλώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μιλήσατε για πολλά θέματα. Απαντήσετε σε συναδέλφους. Εγώ θέλω να επανέλθω σε λίγα θέματα να μην υπάρχουν φραγμοί στη ροή των πληροφοριών ε, που έχει σημασία από το ευρωπαϊκό επίπεδο προς το τοπικό επίπεδο αλλά και από, την, ε, από το ευρωπαϊκό επίπεδο προς ε, όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Θα πρέπει επίσης να δούμε τους φραγμούς στην ψηφιακή αγορά της Ευρώπης που παρεμποδίζουν την διάδοση των μέσων. Μιλήσατε για την πλειάδα των πληροφοριών. Υπάρχει διαφορά μεταξύ πληροφορίας και νέων. Αυτό που είναι σημαντικό για τους δημοσιογράφους δεν είναι κατά ανάγκη το ίδιο σημαντικό για τους πολίτες, τους επιχειρηματίες και τους φοιτητέ. Είπατε ότι θα πρέπει ε, να στέλνουμε το κεντρικό μήνυμα ε, και να κατεβαίνουμε κοντά στον πολίτη. Το 2013 επίσης θα είναι η χρονιά των πολιτών. Καλή ιδέα αλλά μπορεί να μας περιγελάσουν, γιατί εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάθε μέρα, κάθε χρόνο είναι η μέρα των πολιτών. Ε, θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι και οι πολίτες ε, σκέφτονται το ίδιο. Ελπίζω να ενδυναμώσουμε αυτό το συνέστημα στους πολίτες καθημερινά. Για το ρόλο των ΜΜΕ και της επικοινωνία. Είναι σημαντικό να στέλνουμε, να διαδίδονται τα νέα, αλλά υπάρχει και διαφάνεια τα ΜΜΕ ε, διαδίδουν τα νέα, αλλά ελέγχουν και το δικό μας έργο των, ερετών ε, και δημοκρατικά εκλεγμένων αρχόντων. Θα πρέπει να ελέγξουν λοιπόν και το, την εξουσία μας. Σε ό,τι αφορά τα νέα και τους δημοσιογράφους, ε, πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. θα... Δεν έχετε και στην ερώτηση, ναι. Τώρα, θα ήθελα να ενθαρρύνω την εμπλοκή των πολιτών στους σημαντικούς τρόπους για να διαδίδουμε τις πληροφορίες, γιατί αυτό είναι το, ο βασικός αποδέκτης και το κοινό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ανοιχτά δεδομένα, δηλαδή δημόσιες πληροφορίες, ε, και να δίδονται με εύληπτο τρόπο σε πολίτες και σε επιχειρηματίες. Δεν νομίζω ότι κανείς συνειδητοποιεί πόσο πολύτιμες είναι οι πληροφορίες που έχουμε εδώ στα χέρια μας με την ε, βοήθεια των ε, διερμηνέων οι, οι πληροφορίες είναι τόσο σημαντικές που τη χρησιμοποίησε το Facebook ε, για να προσφέρει γλωσσικές υπηρεσίες σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. κοιτάξτε την ημέρα, την ημερίδα ανοιχτών θυρών στις ΗΠΑ Πολιτείες και πώς χρησιμοποιεί η Αμερικανική κυβέρνηση αυτή την ευκαιρία, ευκαιρία αυτή. Ευχαριστούμε η κυρία Τρίπερ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που αναφέρθηκε στην αρχή. Η πολιτικοί είναι αυτή που δημιουργούν μια ιστορία. Και τώρα σε σχέση με χατοφυλάκια και στοιχεία για αυτές τις ε, ευρωεκλογές βλέπω τον ίδιο κίνδυνο να υπάρχει σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν για τα χρόνια αυτής της ε, καινοτόμου δουλειάς ε, και της καινοτομίας. Πολλοί μπορεί κάποιοι να απαντήσουν, α, ήταν για το ένα χρόνο, για το ένα έτος συμβαίνει αυτό και για το άλλο. Λοιπόν, ε, βλέπω να ελοχεύει κίνδυνος εκεί και μετά είπατε στη συνέχεια ότι θα θέλατε να υπάρχει κάποιος τίτλος ε, με θετική απήχηση στη γερμανική Bildzeitung. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι, και αυτή είναι η θέση σας, η πολιτική ήταν, το, ε, ήταν ε, εκείνη που δημιούργησαν το θέμα της κρίσης και σε διαφορά με τον Σαρκοζή ή τον Μπαρόζο η μεγάλα, τα μεγάλα ζητήματα είναι εκείνα που δημιουργούν αυτές τις ιστορίες. Δεν είμαι σίγουρη αν η δική σας προσέγγιση είναι πιστική και δεν κατανοώ το σημείο για τα δίκτυα τα τηλεοπτικά που είπατε. Είπατε δεν υπάρχουν ε, αρκετά χρήματα, μετά είπατε δεν είναι αρκετά αποτελεσματική αυτή η πρωτοβουλία. Ε, θα πρέπει να πάμε στο τοπικό επίπεδο. Γιατί όλοι κάθε φορά, μία φορά τη βδομα... Ε, κάθε εβδομάδα είμαστε στο τοπικό επίπεδο. Η τηλεόραση και αφορά και το διαδίκτυο δεν θα έχουμε αποτέλεσμα στους πολίτες, δεν φτάσουμε τους πολίτες διότι χρειαζόμαστε ένα διαμεσολαβητή μεταξύ των ε, όσων αναφέρονται στα μέσα ενημέρωση, στα μαζικά μέσα ενημέρωση και στα τηλεοπτικά δίκτυα. Δεν ξέρω, αυτά τα οποία είπατε δεν φαίνεται να είναι πολύ πιστικά. Η κυρία Μπαντία, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ και να μας εξηγήσετε όλα αυτά τα θέματα και θα ευχόμουν να έρχεστε πιο συχνά. Στην προηγούμενη εντολή εσείς μας επισκεπτόσαστε περισσότερο, πιο συχνά. Φαντάζομαι και γνωρίζω την ευρύτατο το χαρτοφυλάκιό όσα σήμερα και πρέπει να αντιμετωπίσετε και άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Συμμερίζομαι απόλυτα με όλα όσα είπατε και πολλά από τα πράγματα που αναφέρθηκαν εδώ. Γι' αυτό δεν θα διασπαθήσω περισσότερο χρόνο επ' αυτών. Μόνο μία ερώτηση. Όλες αυτές οι προτάσεις που μας κάνατε, αυτές οι ιδέες που είπα ότι συμμερίζομαι, βασίζονται με τη συμμετοχή, στη συμμετοχή των κρατών μελών που θα δράσουν ως εταίροι. Ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι τα κράτη-μέλη <laughs> με ιδιαίτερη χαρά θα ε, ανταποκρίνονται σε σχέση με τις ανάγκες των, ε, ε, του ευρωπαϊκού επίπεδου. Μας φορτώνουν όλα τα δύσκολα και κρατάνε όλα τα ευχάριστα. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάνιμπαλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε εδώ και μας εξηγήσατε όλα αυτά που ακούσαμε και συγχαρητήρια για αυτή την πολύ περιεκτική έκθεση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να θίξω ε, το θέμα ανάμεσα στη πληροφόρηση και τις ειδήσει. Ε, εδώ ε, έχουμε αυτό που, που λείπει εδώ είναι η είδηση. Αυτά που μιλάμε σε τοπικό επίπεδο νομίζω δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχει εδώ γι' αυτό μιλούσε και ο κύριο Λόκαρτ να υπάρχει κάποιο όραμα, κάποια στρατηγική για το πώς θα κάνουμε συναφές στο ευρωπαϊκό, σε τοπικό επίπεδο, πώς θα βρούμε ιστορίες που θα είναι ενδιαφέρουσες για τα εθνικά μέσα. Αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Ε, δεν θα, έχουμε τη βάση χωρίς την κορυφή και δεν θα έχουμε οποιαδήποτε βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και ξέρω τι εικόνα ε, έχει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να αναπτύξουμε καλές ιστορίες ε, σφαιρικά σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Όπως είπε και ο κύριος Ιβάν, να είμαστε δημιουργικοί και είναι σημαντικό αυτό. Θα ήθελα και πάλι να υποβάλω αυτή την ερώτηση για το όραμα και πώ θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε. Επίσης μια εισήγηση. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σε περιφερειακό επίπεδο. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να συντονίσουμε την Επιτροπή των Περιφερειών, τους τοπικούς, ε, τους τοπικούς βουλευτές, τα τοπικά συμβούλια, στις περιφέρειες και ίσως την Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο ε, ως συντονιστές. Η ανταλλαγή ιδεών και η επεξεργασία αυτών των στρατηγικών στι περιφέρειες είναι χρήσιμο. Αυτό που συμβαίνει στο Λονδίνο διαφέρει πολύ από το τι συμβαίνει σε άλλα μέρη. Ε, τα νέα μέσα νομίζω σιγά σιγά πλησιάζουμε στο στόχο μας αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο το Twitter, τα blogs κλπ. Και τέλος, ε, κάτι το τοπικό πιθανόν είναι αν μιλήσει σε έναν Βρετανό πολίτη για το θέμα του πολίτη, δεν θα δώσουν σημασία. Δεν είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε. Η χρήση της λέξης ε, πολίτης, πολιτότητα, ε, είναι πολύ καλά να τα χρησιμοποιούμε εδώ, αλλά αν ε, πάει κανείς στη Βρετανία και μιλάει για πολίτε, πολίτης, θα, θα, χάσεις το ενδιαφέρον από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να μιλά γι' αυτό. gibt Mimosen in der Europäischen Union. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την ε, ανακοίνωση και για το πρόγραμμα δράσης. Συμφωνώ με όλα όσα λέει. Λείπουν κάποια πράγματα όμως. Πιστεύω. Αυτά που λέτε ενδιαφέρουν αυτούς που ενδιαφέρονται ήδη για την Ευρώπη. Αλλά το 80% των Ευρωπαίων πολιτών δεν ενδιαφέρονται ήδη ή τουλάχιστον ακόμα για την Ευρώπη. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να οργανώσουμε διάφορα γεγονότα και δραστηριότητες με συνέστημα ε, και ενδιαφέρον που θα κάνει τους πολίτες να είναι υπεύθυνοι, ε, περήφανοι που είναι Ευρωπαίοι. 60.000 Βρετανοί που στο Ryder Cup ε, υμνούσαν την Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε τέτοια γεγονότα, παραδείγματο χάρη να διοργανώσουμε κάτι στις Βρυξέλλες και οι τηλεοράσεις θα τα, αναμεταδίδουν αυτά τα γεγονότα, ούτως ώστε ο κόσμος να αισθάνεται περήφανο που είναι Ευρωπαίος. Ε, όταν κάποιος είναι περήφανο που είναι Εβραίος, συγγνώμη, Ευρωπαίος, ε, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι περήφανο που είναι <laughs> Λουξεμβούργιος Έλληνα ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπόρι, παρακαλώ. E, Σας ευχαριστώ. Ένα τέτοιο γεγονός θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πολωνία και Ουκρανία το 2012. Αλλά τώρα σοβαρά συμφωνώ πρέπει να πω με αυτά που η κυρία Επίτροπος μας εξέθεσε σε σχέση με τα νέα μέσα για τη νέα προσέγγιση, για τη νέα αυτή εξειδικευμένη ενημέρωση σε, για όλες τις πρωτοβουλίες, σε εκατοντάδες πρωτοβουλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Έχω μια πρόταση που θα ήθελα να αναφέρω. Σήμερα δεχτήκαμε και υπήρχαν τόσες προτάσεις για πρωτοβουλίες ε, σε σχέση με την πρωτοβουλία για τους Ευρωπαίους πολίτες παράδειγμα. 70% του ευρωπαϊκού δικαίου μεταφέρεται στο επίπεδο των εθνικών νομοθεσιών. Θέλω να πω ότι στα περισσότερα μεγαλύτερα κράτη-μέλη τα μέσα του τύπου, τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε σχέση και με τις ε, εθνικές εθνικές πτυχές ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σημαντικά για να ενημερώνεται ο πολίτης για τα θέματα αυτά ουσίας. Ας σκεφτούμε λοιπόν, ας προβληματιστούμε να συντονίσουμε με τέτοιο τρόπο τα πράγματα ώστε τα ΜΜΕ στα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν για τις πολύ σημαντικές ε, κοινοτικές πρωτοβουλίες των Βρυξελών και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο των Βρυξελών, στις Βρυξέλλες σήμερα. Στα περισσότερα κράτη-μέλη έχουμε πληροφόρηση μόνο για τα αρνητικά τα οποία απορρέουν βγαίνουν από, βγαίνουν από τις Βρυξέλλες ε, ε, και έχουμε αρνητική πληροφόρηση για τις Βρυξέλλες τελικά. Ίσως θα μπορούσαμε να συντονίσουμε έτσι τον ρόλο των ε, κρατικών μέσων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι υπεύθυνα για να ενημερώσουν και για τις θετικές πτυχές που είναι σαν αποτέλεσμα έχουμε ως συμπέρασμα και σαν παρεπόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ εσείς ε, το βρίσκω πραγματικά Πολύ ενδιαφέρον πώς γίνεται λόγος για την ελευθερία του τύπου, για τα θέματα σύνταξης ε, ειδησιογραφίας. Είναι σημαντικό όμως πιστεύω κυρία Ρέντινγκ, εσείς αυτή την προσέγγιση που παρουσιάζετε στο έγγραφό σας, να μεριμνήσουμε να δούμε πώς οι πολίτες συγκεκριμένα μπορούν να είναι οι αποδέκτες αυτών των στοιχείων. Ξέρουμε ότι μειώνεται η αποδοχή για τα ευρωπαϊκά θέματα όταν δεν ε, υπάρχει αυτή, αυτό το στοιχείο. Οι γενναίες, ε, οι πολίτες θεωρούν πολλά πράγματα ως αυτονόητα και καλύτερα περνάνε τα μηνύματα δυστυχώς μέσω των μέσων ενημέρωσης όταν είναι αρνητική ενημέρωση και όχι θετική. Είναι σημαντικό στη στρατηγική μας για την ενημέρωση να είμαστε πιο συντονισμένοι και με καλύτερα διαρθρωμένο τρόπο. Έχουμε μια πλημμυρίδα πληροφοριών που δεν μπορεί να αφομοιώσει και να χωνέψει ο κάθε απλός πολίτης. Κάθε επίτροπος, κάθε γενική διεύθυνση της Επιτροπής, κάθε τμήμα του Κοινοβουλίου, μυριάδες πληροφορίες υπάρχουν και που ναι μεν όλα όλες αξίζουν κάτι αλλά που πολύ δύσκολα εντάσσονται μέσα σε μια σφαιρική πολιτική ενημέρωσης. Το θέμα της αποτελεσματικότητας με την πλημμυρίδα, την χιονοστιβάδα αυτών πληροφοριών που έχουμε δημιουργεί ερωτήματα. Τίθεται και το, διατυπώνεται και το ερώτημα προς εμάς κυρία Επίτροπε. Αυτή τη μάζα πληροφοριών που έχουμε πρέπει να την διηθήσουμε, να την φιλτράρουμε, να δούμε για ποια ομάδα, ποια κατηγορία πολιτών, για ποια χώρα μπορεί κάτι να είναι σημαντικός πληροφορία επικεντρωμένα, με συμπυκνωμένο τρόπο να υπάρξει ενημέρωση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προς τους πολίτες. Με υλικό ενημέρωσης και πληροφόρησης στοχοθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες ως αποδέκτες να μπορέσουν να το αφομοιώσουν αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει πλέον ένα διαφανές πλαίσιο. Υπάρχει εδώ ένας λαβύρινθος. Ε, υπάρχει ας το πω έτσι μια ζούγκλα που ε, με πάρα πολλά ε, δέντρα που δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει μια ε, επισκόπηση του τι συμβαίνει. Και για μένα τίθεται επίσης το ερώτημα, το ζήτημα, πώς η Ευρώπη θα συνδέεται με κάποια πρόσωπα, με κάποια άτομα. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν γι' αυτό. Είπε κάποιος επιτόπου να είναι κανείς παρόν, να είναι γνωστός επιτόπου το πρόσωπό του να μπορεί να το αναγνωρίζει ο πολίτης. Να ξέρει ότι ορίστε αυτός με αυτό το άτομο συμβαίνει το, εξί, το ένα ή το άλλο. Το ίδιο για τους επιτρόπους. Πώς θα βελτιώσουμε αυτά τα πράγματα ώστε οι πολίτες να έχουν έχουν πιο άμεση επαφή από πρώτο χέρι που θα τους διευκολύνουμε. Ο κύριος Ταβάρες παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα κάνω υποδείξεις, όχι ε, ε, ερωτήσεις. Μία γνώμη θα εκφράσω και τρεις ε, συστάσεις. Θέλω να κάνουμε διάκριση δύο ενιών, της προπαγάνδας και της ηθαγένειας. Άκουσα πάρα πολύ καλές ιδέες, καλές για προπαγάνδα αλλά δεν θα πρέπει να μα ενδιαφέρουν ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς είμαστε μια τραγική διαφημιστική εταιρεία, κακή. Η Ευρώπη προσπαθεί να πουλήσει τον εαυτό αυτό της, αλλά μοιάζει ψεύτικη και ο κόσμος δεν, δεν το τρώει, δεν, αγοράζει αυτό το μήνυμα. Ε, τώρα, ε, για να είναι κανείς πολίτης πρέπει να ε, γνωρίζει τα δικαιώματά του. Ε, μόνο όταν γνωρίζει τα χρησιμοποιεί. Και για να τα γνωρίσει μία είναι η ιδέα. Ε, απλούστευση. η Αμερική, η Γαλλία μάλλον, στη Γαλλική Επανάσταση τι έλεγε. Ελευθερία, αδερφοσύνη, ισότητα. Εμείς πρέπει να βρούμε και εμείς το μήνυμά μας, να το πούμε με απλό τρόπο, να είναι ένα είδος συνθήματος. πρέπει να φτάσουμε, ας πούμε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια ιδέα, να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, όχι 27 διαφορετικές. Ε, θα πρέπει να έχουμε, ας πούμε, καταρχάς ε, μια χάρτα δικ, δικαιωμάτων. Έχουμε τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, καλό και απλό έγγραφο, αλλά κατά τα άλλα έχουμε οδηγίες και κανονισμούς που είναι περίπλοκοι. Μιλήσαμε ε, για την προστασία των δεδομένων. Για την προστασία των δεδομένων, ας πούμε, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ω παράδειγμα. Θα πρέπει να έχουμε τι εντολέ για την προστασία των δεδομένων. Δεν θα πρέπει να πουλά τα δεδομένα μου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί χωρί να το γνωρίζω κτλ. κτλ. Εντολέ. Οι Αντίστοιχα με τι 10 εντολέ. Απλούστευση επίση των συμβάσεων περιοδική σφαίρα στο ε, διαδίκτυο. Εκεί που λέει Read our privacy policy. Κάνουμε κλικ και είναι 20-30 σελίδε. Ποιο θα το διαβάσει αυτά. Επομένω, όλοι προσυπογράφουν σε αυτή τη σύμβαση χωρί να διαβάζουν αυτή την πολιτική ιδιωτική σφαίρας. Ε, καλό θα ήταν να απλουστεύσουμε αυτά τα πράγματα με απλά πράγματα, με εικόνες. όταν υπάρχουν ε, οπτικές παραστάσεις, ο κόσμος ε, μπορεί να καταλάβει την πρόκειται χωρίς να χάνει δύο ώρες. Δεν είναι όλοι νομομαθείς, έτσι. Τρίτον, για μας περισσότερο, κάνω έκκληση στους συναδέλφους να πάτε στην ιστοσελίδα Open Congress ε, που τη διαχειρίζεται μία μη κυβερνητική οργάνωση. Ε, είναι μία σύνοψη όλων των ε, νόμων του Αμερικανικού Κογκρέσου όταν συνεδριάζει ή όχι. Μην ασχολείστε με το Facebook και το Twitter κτλ. Γιατί χρειάζεται κανείς ένα χρόνο να το σκεφτεί, ένα χρόνο να το ανεβάσει και μετά εξαφανίζεται. Μην επενδύετε λοιπόν σε αυτά, Facebook, Twitter κτλ. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να υποχρεούται κάθε πακέτο που ολοκληρώνει να έχει μία δέσμη αρχών που μπορεί να τις γράψει κανείς σε μία σελίδα α4, δηλαδή δέκα αρχές ας πούμε. Για τα δικονομικά δικαιώματα ας πούμε, μία σελίδα α4, ε, με λίγα πράγματα. Αυτά, αυτά. Κάποιες... Αυτά είναι κάποιες ιδέες Mange tak, og tak for svaret. Jeg skal være ganske kort. Skal... Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Εν συντομία, όπως κατανόησα την απάντηση, είναι ότι καταφατικά απαντήσατε. Είπατε ναι. Και τώρα τίθεται φυσικά το ερώτημα. Πώς μπορούμε όλα αυτά πιο διεξοδικά να τα πάρουμε, πιο αναλυτικά από αυτό το έγγραφο εργασίας. Μπορεί κανείς να έχει τη μία ή άλλη πρόταση που θα ενταχθεί, μπορεί να υποβληθούν κάποιες προτάσεις, να ενταχθούν κάποιες προτάσεις. Είναι εξαιρετικά αυτά τα οποία προτείνονται. Αυτό το έγγραφο θα το είχαμε λοιπόν ας το πω έτσι, σε αυτές τις διαστάσεις και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ε, με τη δουλειά. Μετά θα ήθελα να αναφέρω ένα άλλο σημείο, πολύ σύντομα, Επίτροπε. Αυτή η πρόταση σε σχέση με τη συνεργασία στον τηλεοπτικό τομέα είναι ένα αρνητικό μήνυμα. Ωραία, γνωρίζω υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, όλοι το κατανοούμε αυτό. Αλλά τώρα ως αιτιολόγηση, ως επιχείρημα αυτής της πρότασης σε σχέση με υφιστάμενους ραδιοφωνικού σταθμούς που αναφέρατε. Υπάρχουν πολλά τέτοια δίκτυα υφιστάμενα δίκτυα και να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, αξίζει αυτό. Σίγουρα κοστίζει. Είναι, ε, υπάρχουν δαπάνες που θα ε, προξενηθούν. Έχει δίκιο η κυρία Τρούπερ σε αυτά που είπε. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι όμως ε, το καταληκτικό σημείο στο οποίο θα ολοκληρώσουμε και θα σταματήσουμε. Πρέπει να προβληματιστούμε να δούμε τι μπορεί περαιτέρω να γίνει. Όπως είπε η κυρία Τρούπερ, πρόκειται για το διαδίκτυο, για παράδειγμα, ραδιο, ε, συγγνώμη, τηλεοπτικές υπηρεσίες που θα μπορούν να παρέχονται και σίγουρα μπορεί αυτό περαιτέρω να αναπτυχθεί και να έχουμε θετικά αποτελέσματα από αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Ρέντινγκ, έχετε τον λόγο τώρα για να απαντήσετε παρακαλώ. Διαφάνεια. Είμαστε τα πιο διαφανή όργανα και η πιο διαφανής ήπειρος στον κόσμο. Έχουμε ένα σώμα ε, τύπου στις Βρυξέλλες όπου μπορούν να υποβληθούν οποιασδήποτε ερωτήσεις, οποιασδήποτε ερωτήσεις. Δημοσιεύουμε τα πάντα, όλα όσα αποφασίζουμε και τα δημοσιεύουμε και σε ε, περιληπτική μορφή. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους βουλευτές που επιθυμούν να επεξεργαστούν αποφάσεις που έχουν ληφθεί στη, στο Γραφείο Δημοσιεύσεων που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και που δημοσιεύει όλα τα επίσημα έγγραφα και τις αποφάσεις δημοσιεύονται επίσης και σύντομες περιλήψεις για τον πολίτη όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται. Άρα δεν χρειάζεται να εφεύρουμε αυτά τα εργαλεία. Ήδη υπάρχουν. Το ερώτημα είναι ποιος κατορθώνει να τα αγγίξει, να έχει πρόσβαση σε αυτά. Και γι' αυτό θέλω να έχω μια μόνο απευθυντική ε, αγορά. Δηλαδή, σαν πολίτης να πηγαίνει κανείς κάπου και να παίρνει απλές απαντήσεις στα ερωτήματά του. Όλα υπάρχουν, είναι στη διάθεση του πολίτη, αλλά πρέπει να είναι κανείς ειδικό για να τα βρει, να, τα, να έχει πρόσβαση σε αυτά. Απλούστευση λοιπόν της πρόσβασης. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Το περιεχόμενο υπάρχει και υπάρχει πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε κανείς να αφομοιώσει. Η συμμετοχή του πολίτη σε όλη αυτή τη συζήτηση τώρα. Μπορώ να σας διηγηθώ πολλές εμπειρίες ε, ε, σε δημόσιους ευρωπαϊκούς χώρους όπου το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν συνεργάζονται και όπου υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε πόλεις, σε περιφέρειες μαζί με τους πολίτες. Αλλά σε αυτούς τους διαλόγους δυστυχώς ε, συμμετέχουν μόνο οι επαΐοντες. Οι άλλοι δεν έρχονται. Και Γι' αυτό θα, ε, έπρεπε, θα μπορούσα να αναφερθώ σε 100 διαφορετικούς τίτλους. Αν ε, στην, στον τύπο έχουμε μόνο τα αρνητικά, τότε δεν θα πετύχουμε ποτέ αυτό που θέλουμε. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω και σας δίνω τα, αποτελέσματα παραδείγματα, πρέπει να έχουμε και τις θετικές επικεφαλής. Όταν στην εφημερίδα Bild, ε, στην πρώτη σελίδα, έχω το 2010 είχα δύο θέματα. Το ένα για την ε, ε, στολιτών δικαιωμάτων και το άλλο για την ισχύουσα νομοθεσία για τα διαζύγια. Δύο επικεφαλίδες στην Bild. Γιατί? Γιατί ήταν κάτι που κατανοούσαν οι πολιτικοί Πρώτον για τα δικαιώματα, λένε α, ε, είναι αυτό το έγγραφο των δικαιωμάτων, μια προειδοποίηση και τώρα έχουμε και τη δική μας προειδοποίηση εδώ στην Ευρώπη, την προειδοποίηση της Reading. Κάτι που σχετίζεται με δύο ε, συγκεκριμένα άτομα. Αλλά είναι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε στην καθημερινή μας δουλειά. Αν θα είμαστε πιστικοί όχι, ε, δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω αυτό. Είναι οι ψηφοφόροι που θα το κρίνουν. Στο τέλος, πρώτα απ' όλα θα νιώθουν ότι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Είναι, τους ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα και θα πάνε να ψηφίσουν. Κατά δεύτερο λόγο, γνωρίζουν για ποιο πράγμα ψηφίζουν. Και είναι δική μας ευθύνη να πετύχουμε αυτά τα δύο θέματα. Και με συζητήσεις σχετικά με το ευρώ δεν θα το πετύχουμε. Λυπάμαι, αλλά το γνωρίζετε. Θα το πετύχουμε με τα δικαιώματα Μιράντα, για παράδειγμα, και θέματα συναφή με αυτά. Θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτά τα θέματα και εσείς θα αποφασίσετε αν είναι πιστικά ή όχι. Το, έτος, το ευρωπαϊκό έτος του πολίτη αξίζει ή δεν αξίζει. Αυτό να σε εσά, διότι τον Μάρτιο θα λάβετε τις προτάσεις μου και αν πιστεύετε ότι δεν αξίζει, τότε θα ψηφίσετε αναλόγως. Είναι απλά δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω. Εγώ προτείνω. Εσείς αποφασίζετε. Άρα, ίσως εσείς να βελτιώσετε αυτά που θα προτείνω εγώ με όλες, τις... τις ιδέες που θα δείτε ή μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι ανοησίες, θα το καταψηφίσετε και το ξεχνάμε. Εγώ το βλέπω ως πρόταση για να συγκεντρωθούμε σε αυτά τα στοιχεία που δεν θα υλοποιηθούν το 2013. Πολλά τα έχουμε ήδη υλοποιήσει το 10 και ε, δεν τα καταψηφίσατε, τα υπερψηφίσατε. Για παράδειγμα, το δικαίωμα στη μετάφραση όταν είναι κανείς σε, σε αστυνομικό σταθμό στο εξωτερικό. Αυτό το υπερψηφίσατε. Είναι στοιχεία τα οποία θα προταθούν. Και ναι, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και ναι, μερικά τουλάχιστον κράτη-μέλη κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Νομίζω σας έχω δώσει κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών. Μάλτα, Ιταλία, Φιλανδία, Σουηδία, Σονία, Βέλγιο, Λετωνία κλπ. Πολύ πολύ συγκεκριμένα προγράμματα και έργα που έχουν υλοποιηθεί στη Σλοβακία. Ε, για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Τρένο πληροφόρηση στη Σλοβενία, ε, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινηματογράφου. Πολλά, πολλές τέτοιες εμπειρίες μαζί με τα κράτη-μέλη που τρέχουν και όταν υπάρχει κάτι θετικό σε ένα κράτος μέλος είναι καλό να το αντιγράψουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συντονίσουμε τις τοπικές στρατηγικές της περιφέρειας, ναι. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών. Πολλές φορές την ξεχνάμε. Ε, ε, ε, έχουν την καλή βούληση, είναι καλή στην επικοινωνία, είναι ερετή από τις περιφέρειες. Ας συνεργαστούμε καλύτερα μαζί τους τις διοργανικές ομάδες εργασίας είναι μαζί μας, συμμετέχουν, είναι όλο δυναμισμό και ενέργεια και ιδέες. Και στην επόμενη μας συνάντηση, κοινή συνάντηση, θα ε, θεσπίσουμε ένα συντονισμένο πρόγραμμα για να συμμετέχουν και εκείνοι ε, στην υλοποίηση αυτών των ιδεών. Δεν έχω άλλη λέξη που να αντικαθιστά τη λέξη πολίτης στη Μεγάλη Βρετανία. Ε, πείτε μου εσείς τι άλλη λέξη θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ε, μερικές φορές μπορεί να είναι και θέμα μετάφρασης, αλλά θα ψάξουμε και θα βρούμε κάποια άλλη λέξη. Συμφωνώ ότι 80% των πολιτών μας δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να τους μιλάμε για την Ευρώπη. Θα πρέπει να τους μιλάμε για τους εαυτούς τους, για τους ιδίους, για τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Ε, για κάτι το οποίο ήταν σκάνδαλο και το οποίο λύσαμε. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προσεγγίσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και των ψηφοφόρων. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και το 20% στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε πιο εκτεταμένες εξηγήσει. Ο αθλητισμός πάντα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο. Έχουμε και τον διαγωνισμό της Eurovision τραγουδιού. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ε, Υπάρχει και το, το βραβείο Λουξ βέβαια, το βραβείο κινηματογράφου. Το βραβείο Λουξ είναι ενδιαφέρουσα ιδέα και θα μπορούσαμε να το ε, εφαρμόσουμε και σε πιο τοπικό επίπεδο. Αν θέλετε τη βοήθειά μου, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό, ε, επειδή αγαπάω πολύ και τον κινηματογράφο, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν είμαι υπέρ της διαφήμισης ούτε της προπαγάνδας φυσικά αλλά υπέρ της αντικειμενικής πληροφόρησης για τις, τις δράσεις μας. Ο τρόπος με τον οποίο εσείς ως μεμονωμένα άτομα και πολιτικοί παρουσιάζετε αυτές τις αντικειμενικές πληροφορίες για να τις κάνετε μη αντικειμενικές, αυτό εναπόκειται στην πολιτική. Εγώ δεν θα μιλήσω για πολιτική. Ε, δίνω αντικειμενικές πληροφορίες για αυτούς που θέλουν να τις μεταδώσουν και να τις αξιοποιήσουν. Το τηλεοπτικό δίκτυο. Υπήρχαν δύο ερωτήσεις για το τηλεοπτικό δίκτυο μετά από μια ανάλυση κόστους ε, φέλους και μια πολύ αντικειμενική ανάλυση θεώρησα ότι είναι πιο υπεύθυνο ε, ε, δεδομένων των κονδυλίων που έχει ο φορολογούμενος να μην συνεχίσουμε με αυτό. Είναι μια απόφαση που έλαβα και ε, εκείνοι που δούλεψαν σε αυτό το θέμα ε, ενημερώθηκαν επισήμως. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι απόλυτα, αλλά είμαστε ευγνώμονε που είχαμε αυτή την ευκαιρία αυτή τη ανταλλαγή απόψεων. Εντάξει. Και πάλι για άλλη μια φορά. Καλά πράγματα κάνουμε και θετικά και πρέπει να μιλάμε για αυτά. Δεν είναι προπαγάνδα. Είναι αναγκαία να, αναγκαίο να μιλάμε, να ξέρουν οι πολίτε γιατί μα ψήφισαν. Δεν μπορούν πάντα να ξέρουν το τι συμβαίνει και γιατί μα ψήφισαν. Έχουμε την κοινή ίδια προσέγγιση. Θα προσπαθήσουμε στου επόμενου ε, μήνε και εβδομάδε και μήνε και χρόνια να φέρουμε πιο πιο κοντά τους πολίτες σε εμά και να βρισκόμαστε μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών και το Συμβούλιο μαζί στην ε, διοργανική ομάδα για την στρατηγική επικοινωνία. Εκεί θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας και να τις συμπτύξουμε και να τις συσφίξουμε ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ. Πολλά πράγματα κάνουμε από κοινού, ίσως πιθανότερο και περισσότερες ιδέες να μπορούμε να υλοποιήσουμε αν κερδίσουμε το Συμβούλιο Συμβούλιο στην πλευρά μα, ω σύμμαχο. Γιατί αν λέγεται «Α, αυτοί οι χασί στις Βρυξέλλες κάνουν ανοησίε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα στι χώρε μα. Πρέπει όλοι να αισθανόμαστε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Και η εθνική πολιτική και το Συμβούλιο όταν πρόκειται για τα παιδιά και τα εγγόνια του. Το θέμα με του τηλεοπτικού σταθμού δεν ρυθμίστηκε προ ικανοποίηση των συναδέφων, αλλά δεν γίνεται τώρα τίποτα άλλο πια. Ίσως να δούμε μια άλλη πρόσθετη εναλλακτική δυνατότητα του χρόνου. Ε, ίσω μπορεί να βρεθεί μια άλλη ιδέα να επιτευχθεί αυτό που ήθελαν οι ευρωβουλευτέ και να υλοποιηθεί έτσι. Με το ραδιόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού ίσω πετυχαίνει. Με το διαδίκτυο να το προσπαθήσουμε. Η κυρία Λόγκαρντ και ο κύριο Σάντε έχουν καθημερινή επαφή με του προσωπικού του υπολογιστέ στο διαδίκτυο. σω μπορεί να γίνει αυτό και να έχουμε με την κυρία Ρέντινγκ μια νέα δυνατότητα έτσι. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Συνεχίζουμε τη δουλειά μα. Περνάμε στο θέμα Ιβαν τώρα. Έτσι, όχι Ιβαν, αλλά εντάξει είναι ο συνάδελφος Ιβαν που θα μιλήσει ε, για το θέμα της ε, Επιτροπής αυτής ε, που είναι αρμόδια για την αηφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013. Κύριε Ιβαν, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί ευθύ εξ αρχή ότι αυτή η Επιτροπή σου θα, θα, θα λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι όταν θα έχουμε μια νέα ε, έκθεση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη συζήτηση αυτή τη στιγμή, προβλήματα τα οποία τον οριζόντια ή κάθετα σχετικά με είτε όλα τα θέματα ή συγκεκριμένα θέματα, αν θα τα συζητά οριζόντια θέματα που και εμείς θα πρέπει να ε, πάρουμε θέση, πρώτα απ' όλα στην Επιτροπή ΣΟΥΡ αναφέρεται η δομή και η ευελιξία του μελλοντικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις διότι αφενός επιθυμείται ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι πιο ευέλικτο. Γνωρίζουμε ότι προβλήματα είχαμε φέτος με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η συνθήκη της Λεσαβόνας στέθηκε σε ισχύ και έφερε νέες αρμοδιότητες στην Ένωση, αλλά το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι αρκετά ευέλικτο για να μας επιτρέπει να κινούμε κονδύλια από τη μια πλευρά στην άλλη και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε αλλά δεν πετυχαίνουμε να βρούμε χρηματοδότηση διότι αυτό το πλαίσιο δεν μας το επιτρέπει. Γι' αυτό υπάρχουν δύο επιλογές στη συζήτηση η μία μια πρόταση για μια δομή με τρία κεφάλαια πολύ μεγάλα που σημαίνει ότι στο πρώτο κεφάλαιο που είναι πολύ μεγάλο ε, τα κονδύλια κινούνται ευκολότερα άρα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία υπάρχει μια άλλη λύση που προτείνει να σκεφτούμε το μελλοντικό πλαίσιο σύμφωνα με την Ατζέντα 2020 δηλαδή να έχουμε τρία μεγάλα κεφάλαια και ε, δύο υποδιακρίσεις. Αν έχουμε ε, διακρίσεις σημαίνει ότι δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι και μπορεί να έχουμε το ίδιο πρόβλημα το οποίο έχουμε και στο ε, τρέχον πλαίσιο. Μια άλλη σημαντική συζήτηση έχει σχέση με τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι μια πρόταση και υπάρχουν ε, συνάδελφοι που πρότειναν όπως το μελλοντικό πλαίσιο να είναι πενταετές έτσι ώστε να συμπίπτει με την ε, θητεία της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου με την ιδέα ότι είναι πιο δημοκρατικό ο καθένας να αποφασίζει για το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο θα είναι δραστήριος δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αν δούμε τις δημοσιονομικές διαδικασίες, διότι οι βουλευτές που θα μελετήσουν το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο ε, αν δεν κερδίσουν στην επόμενη θητεία δεν θα βρίσκονται ε, στην περίοδο που θα λειτουργήσει το πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο θητείε. Υπάρχει άλλη λύση ενός δεκαετούς πλαισίου, αλλά με ε, ενδιάμεση αναθεώρηση, πιο ισχυρή, όπου μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και μια τρίτη λύση, εφταετούς διάρκειας, δηλαδή να διατηρήσουμε το μοντέλο που έχουμε σήμερα. Ένα δημοσιονομικό πλαίσιο με μεγαλύτερη θητεία έχει ε, ένα πλεονέκτημα γιατί οι, πολιτικές, οι ευρωπαϊκές ε, πολιτικές είναι πιο προβλέψιμες, όλοι οι μηχανισμοί υλοποίησης των πολιτικών, αξιολόγησης τους ε, οριμάζουν μέσα σε αυτό το διάστημα και αυτόματα αυτό που αποφασίζουμε είναι πιο αποτελεσματικό και η χρήση των κονδυλίων γίνεται με καλύτερο τρόπο. Τώρα, επειδή διατρέχουμε περίοδο κρίσης και όλα τα κράτη-μέλη και όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι επιφυλακτικά όταν πρόκειται να δώσουν μεγαλύτερα ποσά στο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να είμαστε πιο πιστικοί, να πείθουμε καλύτερα όταν ζητάμε κονδύλια από τα κράτη-μέλη και ε, του ζητάμε να συνεισφέρουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση. και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, ε, Νέων και Αθλητισμού είναι σημαντικό να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν θα ήταν εφικτές αν γινόντουσαν μόνο ανάμεσα σε μερικά κράτη-μέλη δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικές και θα ήταν ε, πιο δαπανηρό για τα κράτη-μέλη να εξετάζουν ατομικά αυτές τις πολιτικές. Δηλαδή, εξοικονομούνται κονδύλια γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται ε, μείωση του κόστους ως αποτέλεσμα. Γι' αυτό σε κάθε πρόγραμμα που έχουμε θα πρέπει να υποστηρίζουμε αυτή την άποψη και να αποδεικνύουμε στα κράτη-μέλη ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον στο πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στα θέματα νέων και αθλητισμού. Πρέπει να διατηρήσουμε τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης που είχαμε και στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, αλλά λέω ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα, αλλά να μην πέσουμε κάτω από τα επίπεδα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχω επισέλθει στις τεχνικές λεπτομέρειες. Αν υπάρχουν ερωτήσεις θα μπορούσα να απαντήσω ίσως αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Την έκθεσή σας για τη 16η Μαρτίου την προβλέπετε και εσείς ε, τον Απρίλιο θα ψηφίσουμε μετά στη συνέχεια. Καταρχήν πρόκειται για τεχνικά θέματα αλλά πρέπει επίσης να προβληματιστούμε και να δούμε ποια είναι τα καλά επιχειρήματα που μπορούμε να βρούμε ώστε να επιχειρηματολογήσουμε και να πούμε ότι τουλάχιστον χρειαζόμαστε αυτά που είχαμε την τελευταία φορά που τότε είχαμε δώσει ήδη σκληρή μάχη. Έχουμε λοιπόν νέα έργα, νέα, νέα καθήκοντα, περισσότερα κονδύλια πρέπει να διατεθούν. Δεν μπορούμε την Κυριακή να έχουμε κατήχηση και να λέμε χρειαζόμαστε το ένα ή άλλο έργο και τη Δευτέρα να μην έχουμε κονδύλια για να επιτελεστεί. Λοιπόν, θα λάβει τον λόγο κυρία και μετά μπορούμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω στη συνέχεια. Παρακαλώ κυρία Τρόιπερ. Θα ήθελα για αυτό το θέμα ως μέλος της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών να πω δύο λόγια. Ο κύριος Ιβαν ανέφερε μόλις τώρα ότι από έξι καθαρούς χορηγούς ε, υπό την ε, καθεδρία του κυρίου ε, Κάμερον στι 16-17 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε ότι επί 10 χρόνια λέει ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό πρέπει να παγώσει. Αν γίνει αυτό πραγματικότητα στο πολιτικό επίπεδο, τώρα με όλα όσα επιθυμούμε να προαγάγουμε δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Τελικό μα συμπέρασμα από όλα αυτά πρέπει να είναι ότι με κανένα τρόπο δεν θα συμβιβαστούμε με αυτό και θα υπάρχει τεράστια αντιπαράθεση με το Συμβούλιο. Σαφώ το Δεκέμβριο με τον προπολογισμό για αυτό το έτο χάσαμε. Αν κάνουμε το ίδιο σφάλμα πάλι δεν χρειάζεται με μεγάλες συζητήσεις εδώ, τότε θα είμαστε θα με σφιχτώ το, σφιγμένο το ζωνάρι ε, γονατισμένοι πλέον, θα γονατιστεί και δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και για το θέμα ποια είναι η πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ω ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να έχουμε καλά θεμέλια. Το πρόγραμμα έρασμο, το πρόγραμμα Κομένιους, το πρόγραμμα των μέσων. Πολλά έχουμε να επιδείξουμε και ξέρω πόσο σκληρά, σκληρή είναι η ε, πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά το γεγονό ότι έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτά τα προγράμματα δημιουργούν ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία Μα κάνει να είμαστε σχετικά ισχυροί. Και αυτά πρέπει επιθετικότατα να τα προωθήσουμε προ τα εμπρό. Έχουμε περισσότερα στα χέρια μα από ότι σε σχέση με άλλα κονδύλια, με άλλε γραμμέ του προϋπολογισμού Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο το οποίο σήμερα το πρωί με εγνώχλησε πολύ και με εξόργησε. Είπε η κυρία Ρέντινγκ ότι στο θέμα της επικοινωνίας για την ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολύ σημαντικό λέει, το θέμα του αθλητισμού για να πετύχουμε να είμαστε κοντά στους πολίτες. Το αντίθετο είπε η Ουγγρική Προεδρία ότι με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές δεν υπάρχουν λέει, κονδύλια για τον αθλητισμό. Αν συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε δύο που ο ένας λέει το ακριβώς αντίθετο του άλλου και από όσα έχουν προαναγγελθεί δεν χρειάζεται να συζητάμε διαμακρών, δεν γίνεται τίποτα και πρέπει πολιτικά να είμαστε πολύ πιο σαφείς στην τοποθέτησή μας και πιο επιθετικοί. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Η διαφορά μεταξύ αυτών που υποτίθεται ότι αναφέρθηκε και αυτών που ακούσαμε από την κυρία Ρέντινγκ είναι πρέπει να πω ε, διαμετρικά αντίθετες οι τοποθετήσεις. Δεν μπορούμε μετά τη Λισαβόνα, τη συνθήκη της Λισαβόνας να έχουμε νέες αρμοδιότητες εμείς να μην έχουμε δυνατότητε και κονδύλια να κάνουμε τίποτα. Αυτογελιοποιούμεθα. Πόσοι αθλητέ είχαν προσέλθει εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, ήδη πριν από τη Λισαβόνα. Και τώρα περιμένουν κάτι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απαράδεκτο αυτό. Είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να πείτε κάτι. Έχετε τον λόγο, Επιτροπή. Παρακαλώ. Ε, let me start. υποστηρίζω τα περισσότερα από αυτά που είπε ο κ. Ιβάν για την ευελιξία, τη διάρκεια και την προστιθέμενη αξία. Ειδικά για την ε, προστιθέμενη αξία, αυτός ο τομέας είναι πολύ σημαντικός και στην προπαρασκευαστική φάση του έργου της Κομισιόν ε, επικεντρωνόμαστε εκεί και όπως είπε η κυρία Τρούπελ, ε, έχουμε καλά επιχειρήματα στον τομέα της εκπαίδευσης, κυρίως εκπαίδευσης αλλά και σε άλλους τομείς. Ο κύριος Ιβαν ζήτησε τουλάχιστον τα ίδια ποσά. Να μην κάνουμε ε, το εξής, το λάθος. Μπορεί η συνολική πίτα να μην αυξηθεί λόγω των πιέσεων από τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να το μοιράσουμε διαφορετικά αυτό το, αυτά τα ποσά που έχουμε, αυτή την πίτα που έχουμε. Δεν μπορώ να προδικάσω τις αποφάσεις ε, του Σώματος των Επιτρόπων. Οι συζητήσεις συνεχίζονται στο εσωτερικό της Επιτροπής, αλλά έχουμε επιχειρήματα τα οποία αναγνωρίζονται είτε εν μέρη είτε πλήρω στην ενδιάμεση έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Υπάρχουν επιχειρήματα για να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα για προγράμματα εκπαιδευτικά. Θα το πιέσουμε από πλευρά Κομισιόν αυτό, αλλά είναι πολύ νωρί ε, για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα η πρόταση θα γίνει στα μέσα, η σχετική πρόταση θα γίνει στα μέσα του 2011 για τον αθλητισμό. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας και δεν ξέρω τι είπε ακριβώς σήμερα το πρωί η κυρία Βασιλείου γιατί δεν ήμουν παρόν. Αλλά αναλύουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε και ποια είναι η προσθεμένη αξία της Ευρώπης στον αθλητισμό. Δεν την έχουμε τελειώσει αυτή την ανάλυση, είναι πολύ νωρί λοιπόν να προδικάσουμε τα συμπεράσματά τη. Όμω να μην ξεχνάμε ότι έχουμε λίγου πόρου, λίγα κονδύλια, άρα θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιε προτεραιότητε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αν η προτεραιότητα θα είναι ο αθλητισμό, αν θα είναι η εκπαίδευση, αν θα είναι κάποιο άλλο τομέα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλου του τομεί. Ίσως αυτό, το, αυτό είπε ακριβώς ε, η κυρία Βασιλείου σήμερα το πρωί. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα εκεί που η Ευρώπη έχει προστιθέμενη αξία. Είναι το μόνο που μπορώ να σας πω προς το παρόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επισημάνω κάτι αν γίνεται. Έχετε εδώ ένα χαρτοφυλάκιο, ένα ε, φάκελο. Κοιτάξτε υπό το σημείο 11. Πάρτε το και αυτό να το βάλετε κάτω από το μαξιλάρι σας, να το θυμόσαστε, να το έχετε. Είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο, ένα έγγραφο εργασίας, εισηγητής ο κύριος Ιβάν όπου τα τεχνικά θέματα απαριθμούνται, αλλά επίσης για όλους που είναι καινούρια μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά θέματα και αυτά που θέλουμε να υπερασπιστούμε μελλοντικά για μας. Οι μόνοι τομείς που έχουμε, Εράσμους Μούντους, πολιτισμός, διαβίου, μάθηση, όλα αυτά απαριθμούνται ένα προς ένα. Και είναι πολύ ευανάγνωστο το κείμενο και εύληπτο και είναι πολύ σημαντικό για τη μελλοντική συζήτηση παίρνει κανεί ε, σημαντικά πράγματα στα χέρια του και δεν τα κοιτάζει πολλέ φορέ. Αυτή τη φορά πρέπει να πω, πάρτε το όλο το 11. Αφαιρέστε το από το φάκελο και βάλτε το στο αρχείο σας. Φυλάξτε το. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο. Θα ψηφίσουμε την επόμενη φορά γι' αυτό. Ο κύριος Ματούλα παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα και εγώ να πιστήσω την προσοχή ε, στο θέμα αυτό, διότι όταν μιλάμε για την ε, περίοδο μετά το 2013, για την στρατηγική 2020, μιλάμε για μείωση των γραμμών, μείωση των κονδυλίων και των διακρίσεων αλλά για μας στο τομέα της, του πολιτισμού και της παιδείας και του αθλητισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει απλούστευση, αλλά αποτελεί και μείζωνα κίνδυνο, διότι τι, εξ, ξαφανίζεται πάντα οι μικρές γραμμές χρηματοδότησης. Εμείς στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα πιο ορατά προγράμματα με ένα πολύ μικρό προπολογισμό, όπως είπατε και εσείς ακριβώς. Έχουμε την γραμμή χρηματοδότηση που είναι μειωμένη, αλλά η ορατότητα είναι πολύ μεγάλη. Και θα ήθελα να ακούσω και εγώ τον κόδωνα του κινδύνου. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Συμφωνώ να μειωθούν όλα αυτά τα κεφάλαια και υποκεφάλαια, αλλά να, να μην εξαφανιστούν αυτό που δεν επιθυμούμε. Για παράδειγμα, ο αθλητισμός γιατί μάταια η συνθήκη της Λισαβόνας έχει εντάξει τον αθλητισμό ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν θα υπάρχει γραμμή του προπολογισμού. Αθλητισμός δεν, δεν σημαίνει μόνο αθλήματα επιδόσεων, σημαίνει και αθλητισμός της βάσης, αθλητισμός ανάμεσα στους νέους και ιδιαίτερα εδώ υπάρχουν αποτελέσματα που δύσκολα καταμετρώνται. Αν το πρωί ο Υπουργό έλεγε ότι μπορεί ένα ευρώ που επενδύεται στον αθλητισμό κάνει εξοικονομήσει των 2 ευρώ, εγώ θα έλεγα ότι ένα ευρώ που επενδύεται στον αθλητισμό των νέων μπορεί να μας δώσει πολύ περισσότερα από δύο ευρώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε καταλάβει αυτό το σημείο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και ευτυχώ έχουμε με το μέρο μας την Επιτροπή προπολογισμών και την είχαμε και στη τελευταία συζήτηση. Θα προσπαθήσουν να πιέσουν το Συμβούλιο για να μας δώσει περισσότερα λεφτά για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Ε, η κυρία Βασιλείου δεν ήταν εδώ σήμερα το πρωί. Η Ουγγρική Προεδρία ήταν και μας είπε ότι η κυρία Βασιλείου ανέφερε χθε ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξουν αθλητικά προγράμματα. Ε, πέστε της λοιπόν, διαμηνήστε της ότι αυτό το θεωρούμε παράδεκτο. Εμείς ε, κάνουμε κάποιες προτάσεις και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να ιτηθούμε εκ των προτέρων. Να μην ξεχάσουμε το έγγραφο εργασία, working document. Είναι εξαιρετικό, πραγματικά το ξαναλέω. Τώρα περνάμε στο θέμα. Ποιο θέμα είναι αυτό τώρα, Τι λέτε, Περνάμε στο θέμα του, ε, της ευρυζωνικότητας, ε, του φάσματος της Έχει ευρυζωνικότητας. Έχεις πολλούς ανεμόμυλους ως αντιπάλους, έχω την εντύπωση. Ε. Πες μας τα σχετικά. Ναι, σας ευχαριστώ θερμά Χαίρομαι πρώτα απ' όλα σίγουρα για το γεγονός ότι τώρα εντωμεταξύ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο σε μια ευρύτερη συζήτηση για αυτά τα θέματα που υποτίθεται ότι είναι πολύ τεχνικά θέματα συζητάμε για αυτά τα θέματα σε ευρύτερο πλαίσιο. Ελπίζω θα συνεισφέρει αυτή η συζήτηση ακριβώς οι πολιτισμικές πτυχές που είναι κάτι που έχουμε ιδιαίτερα κοντά στο πνεύμα και στις προσπάθειές μας στην καρδιά μας θα καταφέρουν να προαχθούν όπου έτσι αξιόπιστα και με σθένος θα αποφασίσουμε, θα εγκρίνουμε μια γνωμοδότηση με προτάσεις ε, που έχουμε στα χέρια μας. Από τη συζήτηση βλέπει κανείς εξόφθαλμα ότι εντωμεταξύ δύο στρατόπεδα ε, ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί το ένα παράλληλα δίπλα στο άλλο. Η μία, το ένα στρατόπεδο λέει τώρα πρέπει να αποφασιστεί να επενδύσουμε στην ευρυζωνικότητα ώστε να είμαστε σε παγκόσμιο πλαίσιο ανταγωνιστικοί. Και γι' αυτό λέει τώρα έχουμε ένα μεγάλο δυναμικό συχνοτήτων που πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι υπάρχουν στοιχεία αριθμητικά πολιτικά για την αντιμετώπιση στενοπών και όλων των άλλων προβλημάτων. Πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι για τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία της πληροφορικής, διότι πολλά άλλα για τη στρατηγική του 2020 δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν αν δεν είμαστε εδώ αποτελεσματικοί. Σίγουρα λυθεύουν κάποια πράγματα εδώ, αλλά επίσης πιστεύω ότι και τα δικά μας επιχειρήματα είναι εξίσου σωστά και σημαντικά. Ότι δηλαδή οι συχνότητες είναι ένα σπανίδι, ε, σπανίζον αγαθό και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στην αντιμετώπιση αντιμετώπιση των συχνοτήτων. Διότι είναι ένα δημόσιο αγαθό οι συχνότητε που ιδιαίτερα για τα πολιτισμικά αγαθά πρέπει να τα εξυπηρετούν και να, τα, να τις χρησιμοποιούμε για να προαχθεί το πολιτισμικό, η πολιτισμική συνιστόσα. Για να το πούμε ξεκάθαρα, εδώ δεν με ενδιαφέρει τόσο το πεδίο των συχνοτήτων μεταξύ 680 MHz και 97 ε, MHz. Ε, Νομίζω είναι ένας τομέας συχνοτήτων όπου στον στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τίθεται αυτό σε χρήση. Ήδη έχουμε πληστηριασμού, δημοπρασίε στη Γερμανία, θα ακολουθήσουν και σε άλλα κράτη-μέλη. Εκείνο που θέλουμε να αποφύγουμε όμω είναι να ανοίξουμε πόρτα και παράθυρο όλε τι πύλε για το άνοιγμα όλων των συχνοτήτων και να έχουμε έτσι μια ενλευκό επιταγή για την χρήση αυτών των συχνοτήτων στο μέλλον. Διότι καταρχήν μόνο προγνώσει και υποσχέσει μα δίνονται για την εκμετάλλευση και χρήση αυτών των συχνοτήτων. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα γίνει και όταν εδώ υπάρχει ας το πω έτσι η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα που σήμερα δεν μπορούμε να κρίνουμε για το μέλλον και ανοίξουμε τις πύλες έτσι για ε, ε, ε, το εύρος κάτω από τα 790 MHz ιδιαίτερα δημοφιλές για τον, την κρατική ραδιοφωνία και τις εκπομπές ραδιοφώνου αυτός δεν είναι, αυτή δεν είναι η σωστή πορεία χρειαζόμαστε ένα πολύ λογικό, ορθολογικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα αποφασίσουμε αν κάποτε η ραδιοφωνία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο ε, να διαθέσει αυτές τις συχνότητες αν κιόλας δεν τις χρειάζεται. Δεν είμαι πρόθυμη με βάση κάποιες απλές προγνώσεις λέει για το μέλλον να ε, κλείσουμε την πορεία προς το μέλλον και να υπονομεύσουμε τα συμφέροντά μας. Όταν ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα για την πληροφόρηση και ενημέρωση στην κοινωνία μας. Να κλείσουμε την ε, πορεία που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αποτελεσματικά προς το μέλλον. Επιπλέον έχουμε και το πρόβλημα των παρεμβολών που ακριβώς ε, υπό το πολιτισμικό πρίσμα δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πριν από την κατακύρωση νέων συχνοτήτων θα πρέπει το θέμα των παρεμβολών και των ε, προβλημάτων να είχε επιληθεί. Τώρα, για την κατακύρωση κάθε συχνότητα, νέα συχνότητα από τα κράτη-μέλη, πρέπει να υπάρξουν όροι και προποθέσει που θα συνδέονται, όπου σαφώ θα προσδιορίζεται ποιο θα παίρνει ποια αντιστάθμιση και ποια αμοιβή, γιατί, για ποια χρήση, ποια συχνότητα και όταν δεν θα χρησιμοποιείται κάποια συχνότητα, τι θα γίνεται. Αυτό θα οδηγήσει στο να, να αντιμετωπιστούν οι δαπάνε ε, των ε, ε, σταθμών με τα, τον εξοπλισμό και τις ε, την υπερβολική επιβάρυνση. Η Βρετανική Αρχή Εποπτείας σε αυτή την περίπτωση νομίζω έδειξε με καλό τρόπο τι πρέπει να γίνει από άλλους και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Μια τέτοια υποχρέωση, όροι και συνθήκες για τα κράτη-μέλη πρέπει να υφίσταται στα κράτη-μέλη πριν από δημοπρασίες και πληστηριασμούς. Ποιος θα υπομίζεται ποιο κόστος, πώς θα επιστρέφεται τέτοιο κόστος, τέτοιες δαπάνες. Αυτό θα ήθελα ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά να το κατοχυρώσουμε. Θα αποφεύγαμε τα αρνητικά την αρνητική αυτή εμπειρία που σημειώνουμε τώρα στη, σημειώνεται στη Γερμανία με εμά. Το ίδιο ισχύει για αυτή την αρχή, η εποπτική αρχή και σε σχέση με τα όσα έχουν δημοσιευθεί ότι όποιος ε, εισάγει προδιαγραφές ETA για αυτές τις συχνότητες ε, έχει τότε σε σχέση με τη λήψη ε, τηλεοπτικών εκπομπών σημαντικές παρεμβολές. Όταν έχουμε καλωδίωση, όταν έχουμε καλωδιακή τηλεόραση και αυτό πάλι εδώ με κάνει να πιστεύω ότι οι πολίτες στα κράτη μας αναμένουν αυτά τα προβλήματα να επιληθούν πιο πριν. Πριν ρυθμίσουμε εμεί κάτι, να προβληματιστούμε να δούμε πώ η επικάλυψη συχνοτήτων και οι παρεμβολέ που θα συνεπάγεται κάποιο τέτοιο πρόβλημα, πώ θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Απλά διαπιστώνουμε εκ των υστέρων ότι υπάρχουν εδώ συχνότητε γειτονικέ ή επικαλυπτόμενε που δημιουργούν τόσο ισχυρέ παρεμβολέ και παράσιτα, τότε τέτοια προβλήματα που δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά μια εκπομπή. Πρέπει λοιπόν να πούμε και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο πριν. Το ότι να, να, αλλάζει κανείς διαρκώς συχνότητες μέχρι να ε, μπορέσει να επιληθεί το πρόβλημα βλέπουμε ότι και σε σχέση με τη στρατιωτική χρήση αλλά και με τους σωστικούς σταθμούς και τη, τη δράση για ε, σωστικά συνεργεία είναι κάτι ιδιαίτερο. Ακούω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλους ότι ήδη τώρα κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είναι σαφές με ποιες εναλλακτικές διαπραγματευτικέ διαπραγματευτικές λύσεις θα καταλήξουμε στην διεθνή διάσκεψη. Μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά παρόλα αυτά μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να δούμε το επανα, ε, αναθεωρημένο πακέτο προτάσεων, την αναθεωρημένη δέσμη ε, για, την, για τα θέματα telecom, των τηλεπικοινωνιών και από πλευράς Ευρωβουλευτών και για μένα και για τους συναδέλφους θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε κάποτε για τις νέες συχνότητες όχι όμω με βάση κάποια αναπόδεικτα στοιχεία και προγνώσει ω ισχυρισμού που λένε να κάνουμε τούτο ή το άλλο. Αν δηλαδή χρειαζόμαστε κάποιε συχνότητε στι ραδιοφωνικέ εκπομπέ, εφόσον αυτά είναι ε, δεδομένα και γνωρίζουμε τι συμβαίνει, δεν μπορεί να ανοίξουμε πόρτα και παράθυρο τι πύλε διάπλατα για τον ανταγωνισμό και την εκμετάλλευση συχνοτήτων χωρί να ξέρουμε ποιο χρειάζεται τι, σε ποιον τομέα και πώ θα κατανεμηθούν, πώ θα επιμεριστούν τι οι quality of service, η ποιότητα των υπηρεσιών, η αναβαθμισμένη ποιότητα πρέπει να είναι γνώμονας. Θέλω σίγουρα να μην τροχοπεδίσω τις εξελίξεις και την πρόοδο, αλλά με τέτοιο πάθος τοποθετούμε με τα επιχειρήματά μου, γιατί το πακέτο μέτρων για τα τηλεπικοινωνιακά θέματα πρέπει να έχει την βέλτιστη αντιστάθμιση μεταξύ κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων σε μια σωστή ισορροπία και έτσι να μπορέσουν να ανοίξουν αγορές αλλά ταυτόχρονα ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να συνεχίσουν να μπορούν να ε, κάνουν εκπομπές ε, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και να μπορεί και η ασύρματη τηλεόραση να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Ό,τι προτείνουμε με βάση τις προτάσεις μου θα πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να πείσουμε την Ήτρε ότι δεν είναι μόνο τα οικονομικά επιχειρήματα που έχουν σπουδαιότητα και διαδραματίζουν ένα ρόλο αλλά και η πολυμορφία του τύπου, ο πλουραλισμός ε, της ενημέρωση, όλα αυτά και τα πολιτισμικά είναι αξίες. Σας ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Πέτρα για την πολύ καλή συνεργασία ε, κατά το παρελθόν πριν από την εκπόνηση αυτού του θέματος. Πολύ καλά και με τους σκιώδεις εισηγητές ε, στην Επιτροπή ε, Πολιτισμού είχε συνεργαστεί και χαίρομαι ε, εδώ και γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την καλή θετική συνεργασία. Μπορώ να συμφωνήσω με τα περισσότερα που ανέφερε η Πέτρα πιο πριν, διότι πιστεύω, θεωρώ ότι δεν βρισκόμαστε σε αντίθεση μεταξύ πολιτισμικών συμφερόντων συμφερόντων και οικονομικών συμφερόντων. Πάλι εδώ, σε σχέση με τη συζήτηση με την Ήτρε, πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη για τον ραδιοφωνικό τομέα, για παράδειγμα, και τι οικονομικέ επιπτώσει που διαμορφώνονται και το μεγάλο υψηλό δυναμικό οικονομικό που υπάρχει. Μεγάλο αριθμό ε, των όσων απασχολούνται στην δημιουργική ε, παραγωγή τέτοιων εκπομπών πρέπει να μα κάνει να διασφαλίσουμε αυτό τον τομέα. Να μην πούμε είναι ένα δεινόσαυρο, είναι κάτι ανεδαφικό και παροχημένο περιεχομένου που πρέπει να πεταχθεί στα σκουπίδια ή να τεθεί στο αρχείο και ιδιαίτερα σε σχέση με την τηλεόραση, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους broadcaster, τους παρόχους δείχνει ότι είναι μια αγορά που έχει ε, δυναμικό και πρέπει αυτές οι πτυχές ε, με, τα, με τον καλύτερο τρόπο, με τα σωστότερα επιχειρήματα να προχωρήσουν. Εδώ θα ήθελα μια πτυχή να τονίσω, μια βελτίωση της ε, κάλυψης του χώρου της υπαίθρου και αυτό είναι σημαντικό για μένα και θέλω να επισημάνω ότι ακριβώς η πρόσβαση η προσπελασιμότητα στο εύρος, στο ευρυζωνικό φάσμα πρέπει να συνδέεται όσον αφορά τις συχνότητες ότι ακριβώς κάποια ανάπτυξη πρέπει να διασφαλιστεί για το χώρο της υπαίθρου. Το θεωρώ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θέσουμε όρους και προϋποθέσεις ώστε να διασφαλίσετε ότι όλα αυτά τα οποία θα αφορούν την απελευθέρωση συχνοτήτων να εμπλέκουν και τις περιφέρειες και το χώρο της υπαίθρου. Να υπάρχει το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο πρόσβασης στα ευρυζωνικά για τους πολίτες της Ευρώπης και το διαδίκτυο. Έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την Ήπεθρο. Υποστηρίζω και το θέμα το οποίο ανέφερε η Πέτρα, το θέμα των παρεμβολών δηλαδή και των παρασίτων, ε, ε, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων. Να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Να μην πούμε επειδή τώρα έχουμε το 800, ε, την 800η συχνότητα που απελευθερώνεται, λύθηκαν τα προβλήματα. Μόνο και με αυτό. Πρέπει πάντα τα προβλήματα με τις παρεμβολές να τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό βρίσκεται στη φύση, έγκυται στη φύση αυτού του φάσματος ευρυζωνικότητας και με την πρόοδο της ε, τεχνολογίας ή τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα να τις χρησιμοποιήσουμε πριν όμως ε, μετατεθούν ή ε, πολιθούν συχνότητες, ε, δημοπρατηθούν και κυρίως ποιος θα υπομειστεί όλα τα κόστη στη συνέχεια αν όλα αυτά γίνουν πρωτού, ρυθμιστούν αυτά όπως πρέπει και με τους παρόχους για τις διευρυμένες δυνατότητες δυνατότητες εκμετάλλευσης αυτών των συχνοτήτων, αυτοί αποκομίζουν το όφελος. Στο τέλος όμως η επιβάρηση για την απελευθέρωση των συχνοτήτων επιβαρύνει τους Δήμους, τις κοινότητες, διότι σε όλους τους χώρους εκδηλώσεων για παράδειγμα, όταν έχουμε ραδιοφωνικές ε, ε, μεταδόσεις, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά συνεπάγονται έξτρα ε, επιπλέον κόστος και δαπάνες για να αντιμετωπιστούν παρεμβολές, παράστα κτλ. Βλέπουμε εδώ σε σχέση με την καλωδίωση έχει, ποια είναι τα μειονεκτήματα. Στο τέλος τέλος επιβαρύνεται το καταναλωτής να αγοράσει νέες, τηλε, νέες ε, συσκευές ε, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ε, εδώ τίθεται το πρόβλημα ποια είναι η πρόσθετη αξία που δημιουργούμε, ποιο είναι το κέρδος και ποιος θα υπομειστεί το κέρδος και ποιος την επιβάρυνση. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει πιο πριν, εκ προημίου, να έχουν πολιθεί. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο και να αποφασίσουμε τη διεύρυνση των συχνοτήτων πριν ρυθμίσουμε όρους και προϋποθέσεις και απελευθερώσουμε κάτω και από τη συχνότητα των 790 τα πάντα, πρέπει πρώτα να κάνουμε τη δουλειά μας στο επίπεδο των 800 όσον αφορά τη συχνότητα και μετά να δούμε τις άλλες δυνατότητες. Το όφελο το ψηφιακό το οποίο μπορεί να αποκομιστεί όταν διεξάγεται αυτή η συζήτηση, σε κάποιες χώρες δεν έχουμε υλοποιήσει καν όλα αυτά. Έχουμε σε κάποιες σε 17 χώρες ε, δεν έχουμε ψηφιακή τηλεόραση, αλλά έχουμε την παλαιού τύπου ακόμα τηλεόραση στις εκπομπές Βρισκόμαστε πίσω λοιπόν σε πολλά σημεία. Πρέπει πρώτα να κάνουμε σωστά τη δουλειά μα πριν υιοθετηθεί μια για όλους γενική ρύθμιση. Και τώρα όσον αφορά την Σύνοδο κορυφής για τις συχνότητε και τον επιμερισμό πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό σε σχέση εκτό ε, από τις συχνότητε ε, μέχρι 800, 800 MHz πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατό να προχωρήσουμε χωρίς να ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις. Τώρα αν θα έχουμε μετά το 2016 μια εναλλακτική διαπραγματευτική δυνατότητα για να ξανασυζητήσουμε το θέμα και να το διαπραγματευτούμε, θα το δούμε αυτό. Σήμερα όμως πρέπει να καθοριστούν όλα αυτά. Μέχρι το 2012 να πούμε το τι μπορεί να γίνει εντάξει. Αν θα πρέπει να δούμε κάποιες ε, τεχνικές εξελίξεις το 2016 να τις συζητήσουμε. Όμως η συζήτηση δεν σημαίνει άνοιγμα όλων των εναλλακτικών δυνατοτήτων, ότι αυτό θα γίνει τελεσίδικα τότε. Το ένα βήμα προσεκτικά μετά το άλλο πρέπει να ακολουθήσει. Αυτό δεν περιορίζει, δεν θα περιορίζει τις εναλλακτικέ εναλλακτικές δυνατότητες διότι αν είχαμε ας το πω έτσι ήδη αυτή τη δυνατότητα ενώπιόν μας θα είχαμε κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Πρέπει να δούμε αν η βιομηχανία, οι κύκλοι της επικοινωνίας μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις δυνατότητες που τους προσφέρουμε. Δεν είναι απεριόριστο αυτό το αγαθό. είναι πεπερασμένο και αν μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση win-win ε, ε που θα είναι κερδοφόρα για Στι πλευρέ, πλευρές, ε, τότε αυτό θα είναι το πιο θετικό. Αλλά σε αυτό το σημείο σίγουρα μπορούμε να δημιουργήσουμε κατάσταση όπου η πρόσθετη αξία θα δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για του πολίτε μα. Και αυτό θα είναι σημαντικό ακόμα και όταν θα έχουμε θέματα επιμερισμού. Θα χαιρόμουν έναντι τη Επιτροπή Ήτρα και για την ακρόαση αυτή και τα επιχειρήματα που έχουν ε, ακόμα μ, πιο ξεκάθαρα διαμορφωθεί και ε, ανάγλυφα παρουσιαστεί να ληφθούν υπόψη. Διαπραγματευθήκαμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα για να πετύχουμε τη δέσμη μέτρων για τι τηλεπικοινωνίε. Μετά από σκληρέ διαπραγματεύσει καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Αυτά τα συμπεράσματα δεν πρέπει να τα πετάξουμε στην κάλαθο των αχρήστων, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για το σημερινό, το, το επόμενο έγγραφο για την πολιτική, για το φάσμα τη ευρυζωνικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξουν αυτό το αίτημα οι συνάδελφοι τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Σα ευχαριστώ, λέγει Πρόεδρο. Χαίρομαι ότι οι δύο σα έχετε την ίδια άποψη. Αν από κοινού συνεχίσουμε τι προσπάθειε, θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σάκε νομίζω έχετε να πείτε κάτι διαφορετικό πιστεύω. Ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, τους συναδέλφους. Ήταν ε, επικοδομητική διαδικασία ε, δεδομένου του περίπλοκου του χαρακτήρα του, θε... χαρακτήρα του θέματος, τεχνικού χαρακτήρα του θέματος. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις και κάποια θέματα που ήθελα να θίξω τα κάλυψαν άλλοι συνάδελφοι. Αυτό που προτείνει η Κομισιόν είναι να αξιολογήσουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Όταν καταρτίζουμε πολιτικές για τις τεχνολογίες, η πρόκληση είναι να το κάνουμε γρήγορα όταν υπάρχουν τεχνολογίες και προσεκτική για να σεβαστούμε τις μεταβάσεις, τα βήματα μετάβασης. Αυτή η ευελιξία θα πρέπει να αναζητηθεί και να τονιστεί Διερωτώ με Φερρυπίν γιατί προτείνεται η τροπολογία 8, γιατί υπάρχουν ε, δια νόμου Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, για θέματα ευρυζωνικότητας και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών και της κατάστασής τους. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τρόπου που η ραδιοτηλεόραση, οι τηλεπικοινωνίες και τα διάφορα δίκτυα λειτουργούν στις διάφορες χώρες μέλη λόγω διαφορετικής φύσης. Ε, θα πρέπει να έχουμε ίδια πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αξιολογούμε σωστά και αντικειμενικά και να μην αφήνουμε τα συμφέροντα των κρατών μελών να επηρεάζουν την αξιολόγηση, ούτω ώστε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα του τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έπειτα να εξασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ε, εκπροσωπούνται στην παγκόσμια σκηνή. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει την τροπολογία 8. Κυρίως στο τελευταίο τμήμα όπου διαγράφηκε ένα τμήμα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Η εναλλακτική τότε είναι ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Γιατί δεν θέλουμε δηλαδή μια κάποια εναρμόνιση, ούτω ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Άρα ένα ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι βασικές μου ερωτήσεις. Ως προς τα υπόλοιπα, καλύφθηκα. Θα ξανακοιτάξω την έκθεση και θα προτείνω και κάποιες τροπολογίες. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ από την Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας των Πληροφοριών και της Ενημέρωσης. Άκουσα λιγάκι την παρέμβαση της κυρίας Ρέντινγκ στο τέλος και την συζήτηση για τον προϋπολογισμό και βλέπω ότι πολλά θέματα ο Επίτροπός μου και η Γενική μου Διεύθυνση θα πρέπει να τα παρακολουθήσουν εκ του σύνεκης, άρα να εμπλακούν στο έργο της Επιτροπής σας. Πέρα από την ψηφιοποίηση με την Ευρωπαϊκή, πολλά πράγματα που κάνουμε για το περιεχόμενο και το media, το Εράσμους για τους ε, δημοσιογράφους, ε, το ρόλο της ε, νεολαίας στην κοινωνία των, των πληροφοριών και της επικοινωνίας. Κάνουμε πολλά, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις συνέργειες, ούτως ώστε οι αξίες αυτής της Επιτροπής σας ε, ενσωματώνονται στο πρόγραμμα εργασίας μας. Θα ήθελα να κάνω 4-5 σύντομα σχόλια, απαντώντας ε, στα όσα ακούστηκαν. Καταρχάς, είναι σημαντικό η πρότασή μας για το φάσμα να συζητηθεί σε πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γιατί είναι μια πρόταση όπου είναι κεφαλιό του σημασίας ε, ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ε, για να δούμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε το δημόσιο αγαθό αυτό και πώς θα διαχειριστούμε το πολύτιμο αυτό αλλά ε, πεπερασμένο αγαθό. Πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό το αγαθό. Υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία, η ανακούφιση από τις φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα δούμε ε, μέσα σε ένα, σε ένα πλαίσιο και να τα αντισταθμίζουμε, να αντισταθμίσουμε τα μεν και τα δε, να δούμε τι παζάρια μπορούν να γίνουν, ε, τι συνεσταμένες μπορούμε να βγάλουμε και ανάλογως θα κάνουμε και τις προτάσεις μας. Η επίπτωση στον πολιτισμό είναι το δεύτερο σχόλιο. Θα ήθελα να πω εν παρόδο ότι ο πολιτισμός είναι ένα ευρύτατο θέμα. Δεν είναι μόνο το ότι κερδίζουμε από τις ιδιωτικές και δημόσιες, από την ιδιωτική και δημόσια Ε, ο πολιτισμός δεν είναι δωρεάν. Μην ξεχνάμε την επίπτωση του πολιτισμού ε, εν το συνόλο του. Και όχι να δούμε τα συμφέροντα ενός τομέα και μόνο. Αν κοιτάξουμε τα συμφέροντα τώρα ενός τομέα, συμφωνώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ραδιοτηλεόραση θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Δεδομένου όμως το, το ότι το φάσμα για το οποίο μιλάμε είναι ένα μικρό τμήμα του φάσματος, αν συμφωνήσετε με την πρόταση της Κομισιόν, μπορούν τα μέσα ή τα κανάλια, ραδιοτηλεόραση λοιπά να έχουν ε, από τετραπλάσια στους δεκαπλάσια κανάλια. Επίσης, τι θα γίνει ε, για τη μετάβαση στην τρισδιάστατη ε, high definition τηλεόραση. μπορούμε στο μέλλον να έχουμε τόσα πολλά κανάλια όσο και σήμερα. Ε, και καθένα να είναι τέλειο, να είναι όπως πρέπει. Αυτό που προτείνουμε ε, δεν νομίζω ότι απειλεί το μέλλον της ε, ραδιοτηλεόρασης. Δεν θέλουμε να απειλήσουμε το δυναμικό και το μέλλον της ραδιοτηλεόρασης. Τώρα, για το μέλλον, για το θέμα του μέλλοντος. Άκουσα τους ε, προηγούμενους ομιλητές ότι συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για το μέλλον μέχρι να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία. Εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε μια πρόταση για το μέλλον και κάποιες από τις απολογές, οι 7 και οι 20 όμως, μας ζητάνε να προδικάσουμε το μέλλον. Για τις παρεμβολές που ανέφερε η συγγήτρια, πολύ σωστά, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα των κινδύνων από τις παρεμβολές και να ε, επιτρέψουμε την αποσημείωση. Ε, δεν ξέρω τώρα αν τα κράτη-μέλη θέλουν η Ευρώπη να επιτρέψει αποζημιώσεις. Πάντως, ε, εκείνος που ζητάει τις αλλαγές, αν χρειάζονται και αποδειχθεί ότι χρειάζονται αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να προβλεφθούν και οι αποζημιώσεις. Τώρα για τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις, τα LTE κτλ. θα πρέπει να υπάρξουν ε, πρότυπα, τεχνολογίες ούτως ώστε να μειωθούν τα προβλήματα εγκαίρως. Υπάρχει ήδη πρόοδος και για τα μικρόφωνα και για τα LTE. Τα δύο τελευταία σχόλια για την ταχύτητα και τη διατήρηση των εργαλείων για να δημιουργήσουμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε μια ικανοποιητική ταχύτητα. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το δυναμισμό της ραδιοτηλεόρασης, αλλά και για τους υπόλοιπους δυνητικούς χρήστες του φάσματος, από ό,τι ενημερωνόμαστε, ίσως τα μισά κράτη-μέλη χρησιμοποιούν και αναλογικά και ψηφιακά στοιχεία. Ε, η Ιρλανδία, η Πολωνία, α, από το 2012 κάπου θα μείνουν ουραγοί. 2013, συγγνώμη. Το θέμα είναι όμως ότι όλοι οι, operator, οι operator παντού να, πρέπει να, να μπορούν να έχουν καθαρό σήμα. Επίσης, ένας κοινό κατάλογος θα είναι αντικειμενικός. Μια κοινή φωνή από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο πολύ κρίσιμα πράγματα και χαίρομαι, κυρία Σάκη, που το τονίσατε. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που προάγουν αυτές τις αρχές. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συλλογικά θεωρούν ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα που ενσωματώνουν την σημασία της πρότασης της Κομισιόν. Και ελπίζουμε αυτή το τομείς να προταχθούν περισσότερο. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτές τις αξίες ε, προάγει η Κομισιόν. Μία σύντομη επερώτηση σε αυτά που είπε ο κύριος Μαντλέον σε σχέση με το ε, αναπτυξιακό δυναμικό, σε σχέση με την τρισδιάστατη τηλεόραση, ότι όλα αυτά διασφαλίζονται μέσα στο πλαίσιο των σημερινών διάβλων, των σημερινών κατα... καναλιών ή πέρα από αυτό. Νέα προγράμματα θα μπορέσουν να δημιουργηθούν ώστε νέοι πάροχοι να μπορέσουν, να το πω έτσι, να εμπλακούν στην διευρυμένη αγορά, στον ανταγωνισμό. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτά τα οποία είπατε ή όχι. Το θέμα είναι ποιες τεχνικές ε, δυνατότητες ε, του δυναμικού, τεχνολογικού δυναμικού στο ευρυζωνικό φάσμα είναι εφικτές. Ποιες τέτοιες δυνατότητες είναι ε, εφικτές, ποιες νέες μορφές θα υπάρξουν, θα υπάρξουν νέα κανάλια. Όλα αυτά τα, όλο αυτό το δυναμικό δεν έχει σήμερα, δεν το έχουμε σήμερα εκμεταλλευτεί. Υπάρχει επαρκές περιθώριο, επαρκές πλαίσιο. Μήπως δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε για το διαδίκτυο τι θα γίνει προτού ξεκινήσουμε και μας πούν πρώτα τεχνική τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματική ε, εναλλακτική λύση στον τομέα των επικοινωνιών και του ευρυζωνικού φάσματος. Και όταν θα τα έχουμε ρυθμίσει αυτά τότε θα πρέπει να δούμε για αυτές τις συχνότητες και ο τομέας της τηλεπικοινωνίας να ληφθεί υπόψη, ώστε να έχουμε την ε, πιο αποτελεσματική χρήση των συχνοτήτων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών πρώτα. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικό θέμα. Τα νούμερα που σας έδωσα είναι μια απόπειρα να κάνουμε προσωμείωση ε, στο μέλλον ε, για την εξέλιξη του φάσματος με τη σημερινή τεχνολογία. Δηλαδή κάνουμε κάποιες ε, υποθέσεις, συντηρητικές υποθέσεις. Η μία από αυτές είναι ότι πάντα θα χρειαζόμαστε ε, το ίδιο βαθμό φάσματος για να έχουμε τρισδιάστατη υψηλής ευκρίνειας τηλεόραση. Δεύτερον, αυτό που λέμε σήμερα τρισδιάστατη ραδιοτηλεόραση, σε καμία χώρα δεν θα προσφέρεται ευρυζωνικά. Σήμερα ε, υπάρχει ένα μείγμα τηλεόρασης IP. Και το φάσμα που θα υπάρχει στη διαθεσή μας μετά τις προτάσεις της Κομισιόν θα επιτρέπουν σε κάθε κανάλι που εκπέμπει σήμερα, σε οποιαδήποτε μορφή αναλογική, ε, ψηφιακή ε, ε, η υψηλής ευκρίνειας να εκπέμπεται ε, τρισδιάστατα HD, δηλαδή με υψηλή ευκρίνεια. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα κανάλια θα υπάρχουν παράλληλα. Το θέμα είναι να δείξουμε πόσο χώρος υπάρχει με τις σημερινές τεχνολογίες. Και συμφωνώ αυτό που υπόθηκε, ότι και οι τεχνολογίες της τηλεόρασης και άλλες, οι άλλες ευρυζωνικές τεχνολογίες θα γίνονται όλο και πιο απλές, δηλαδή θα χρειάζονται όλο και λιγότερο φάσμα να καταναλώνουν. Και δεν θα παίρνουμε δηλαδή το ψωμί του ενός τομέα για να το δίνουμε στο, στον άλλο. Αν επιταχυνθούν οι τεχνολογικές ε, εξελίξεις, οι τεχνικοί θα πρέπει να εξετάσουν πολύ πιο συχνά το πώς οι τεχνολογικές αλλαγές και τα επιχειρηματικά μοντέλα μας οδηγούν στην προσαρμογή των ορίων ανάμεσα στους διαφορετικούς τομείς. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα. Γιατί δεν περιμένει κανένας όλη τη τηλεόραση να γίνει τρισδιάστατη την επαύριο. Φυσικά αυτό το θέλουμε. Αν όλα γίνουν ε, δυσδιάστατα και υψηλή ευκρίνεια, μετά την εφαρμογή τη πρόταση τη Κομισιόν θα έχουμε, μπορούμε να έχουμε τετραπλάσια κανάλια. Μάλιστα, ευχαριστώ. Βλέπει κανεί ήδη τώρα κάπω από αυτέ τι τοποθετήσει που ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι λένε μάλλον πιθανότατα ίσως μπορεί να γίνει. Έχουμε λοιπόν ισχυρισμούς ε, και υποθέσεις. Ξέρουμε ότι η τεχνολογία θα εξελιχθεί και πιθανόν στο μέλλον δεν θα χρειάζονται οι ραδιοφωνικές εκπομπές τόσες πολλές συχνότητες όσο όσες σήμερα. Βρισκόμαστε αυτό το, αυτή τη στιγμή στο επίπεδο υποθέσεων εργασίας για το μέλλον. Καλό θα ήταν λοιπόν πρώτα να μεριμνήσουμε και να δούμε τι θα γίνει με τα 800 ως συχνότητα και τι θα γίνει με τις τεχνικές, τεχνολογικές εξελίξεις πώς θα αντιμετωπιστούν τα παράσιτα, οι παρεμβολές. Διότι και εδώ έχουμε το πρόβλημα. Αν μιλάει κανείς με διαφορετικούς τεχνικούς επαΐοντες, παίρνει από κάθε ένα διαφορετική απάντηση για τα διαφορετικά αυτά θέματα. Ας πάρουμε τα βέβαια και ας αφήσουμε τις υποθέσεις. Πολλά εξαρτώνται αν κάνει λόγο κανείς με, ε, για αυτά τα θέματα ε, με ένα ε, τεχνικό επαΐοντα από τον τομέα των ραδιοφωνικών εκπομπών ή των, με των τηλεπικοινωνιών. Ο καθένας έχει διαφορετική κοσμοθεωρία και διαφορετικές απόψει και θεωρίες. Από διαφορετικές υποθέσεις ξεκινάνε για το τι χρειάζονται οι τηλεπικοινωνίες και οι εκπομπές. Πρέπει πρώτα να βρούμε μια κοινή γλώσσα. Αυτό το έμαθα τώρα σχετικά πρόσφατα. Ξέρουμε επίσης ότι για πολλά πράγματα κάνουμε λόγο όπου δεν γνωρίζουμε ακριβώς, επακριβώς τι συμβαίνει και από τις επιχειρήσεις τις ίδιες παίρνουμε και κάποιες αξιοπερίεργες απαντήσεις. Αφενός μας λένε στις Βρυξέλλες χρειαζόμαστε λέει πολύ περισσότερο χώρο χώρο για συχνότητε, όσον αφορά τι ίδιε συχνότητε, Ολόκληρους όγκου συχνοτήτων. Στην Γερμανία, στην ε, Σύνοδο για τα Μέσα ενημέρωση, μου είπανε ότι η ίδια επιχείρηση καλωδιακών λέει «Μα γιατί να καταργήσουμε τη δυνατότητα αυτή, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, έχουμε αρκετό χώρο, αρκετέ συχνότητε, στα καλωδιακά ήδη σήμερα». Και κάποτε λέει ο πολιτικό, ε τι θα γίνει, ποιον θα πιστέψω από όλου αυτού που μου λέει ο ένα το α, ο άλλο το ω, τα πιο αντίθετα πράγματα. Α αφήσουμε να δούμε τι γίνεται με συχνότητα των 800, α επιληθούν τα τεχνικά προβλήματα πρώτα, α μεριμνήσουμε τα φάσματα τη ευρυζωνικότητα που υπάρχουν στη διάθεσή μα να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και ελέγξιμα από όλου μα και να δούμε μετά ποια πορεία θα ακολουθήσουν οι εξελίξει και να δούμε αν χρειάζεται η απελευθέρωση άλλων συχνοτήτων για ποιο σκοπό και πώ. Δεν πρέπει σήμερα να καθοριστούν τελεσίδικα και καθοριστικά αυτά, να μην ανοίξουμε πόρτα παράθυρο και πύλε για όλες τις εξελίξεις ανεξέλεγκτα, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται τώρα να προδικάσουμε το τι θα γίνει στο μέλλον και έτσι να μην έχουμε δυνατότητε πλέον στο μέλλον να κάνουμε κάτι λογικό. Ίσως δύο λόγια σύντομα για την ερώτηση της κυρίας Σάκε, την παρέμβασή της. Το πακέτο μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες λέει με σαφήνεια ότι τα κράτη-μέλη έχουν αρμοδιότητα επ' αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί σε αυτό το έγγραφο να αποδυναμώσει έντονα αυτή την τοποθέτηση και να πει δική μου είναι η αρμοδιότητα για τα θέματα συχνοτήτων. Δική μου ως, επιτροπής, ως Επιτροπή. Αυτό είναι το σημείο που με την τροπολογία 8 προσπαθώ να ανακτήσουμε το έδαφος εμείς. Και πάλι για το πακέτο μέτρων για τα τηλεπικοινωνιακά να είναι τα κράτη-μέλη τα αρμόδια. Το ότι ίσως σε τέτοιου είδους διασκέψεις όταν έχει κανείς 27 ε, κράτη-μέλη ότι ε, θα είναι δυνατόν ε, να υπάρξει, να ρυθμιστεί το θέμα των τοποθετήσεων, πώς θα υπάρχει μια ενιαία θέση, είναι σαφές, σαφώς θέμα εντολής που πρέπει να δοθεί ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνη της να καθορίζει τις προτάσεις. Πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί μέσα στο πακέτο για τα τηλεπικοινωνιακά που θα ρυθμίσουν αυτά τα θέματα. Γιατί οι θέσεις των κρατών μελών για τις συχνότητες είναι τόσο διαφορετικές και τις συχνότητες τις εκμεταλλεύονται τα κράτη-μέλη ήδη τόσο διαφορετικά που ήδη στις μεθοριακές περιοχές, στις συνοριακές περιοχές έχουμε πολλά προβλήματα με παρεμβολές, παράστα κτλ. Πιστεύω με αυτή την πολιτισμική ε, πολυμορφία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σκόπιμο να ρυθμίζει τα πάντα για τα 27 κράτη-μέλη. Εδώ θέλουμε τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τις ανακτήσουμε κάπως και να διαμορφωθεί το πακέτο μέτρων για την τηλεπικοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγει η Πρόεδρος, ευχαριστούμε την εισηγήτρια, σκιώδη εισηγήτρια επίσης. Θα είναι δυσχερής η πορεία προς το μέλλον. Και επειδή και στην Ευρωβουλή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το ξέρετε αυτό κύριε Μαντλέν, αλλά Πιστέψτε με, πιστέψτε μας, προσπαθούμε παρόλα αυτά οι απόψεις μας να μπορέσουν να συγκλίνουν και κάπως να είναι τέτοιου είδους ώστε να τύχουν πλειοψηφία. Θα μεριμνήσουμε να υπάρξει πλειοψηφική τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε θερμά. Είναι καλό και θετικό το θέμα αυτό της εκπροσώπησης των 27 κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Είναι ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό το θέμα σίγουρα όπως και στην διάσκεψη για την UNESCO αντιμετωπιστή δεν έχω καμία αντίρρηση. Γιατί τότε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν εκείνη που ως προπομπός, ως πρωτοπόρος προχώρησε και πέρασαν αυτά τα αιτήματα. Ελπίζω ότι αυτά ως προτάσεις ε, διατυπώσατε και με την θετική, τις θετικές παρατηρήσεις ή επικρίσεις που έγιναν από πλευράς μας θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 2 Φεβρουαρίου, όχι, στις 3 Φεβρουαρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία που εκπνέει για την κατάθεση τροπολογιών για αυτό το έγγραφο της κυρίας Καμα Έμπερτ. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν παρούσα για αυτό το θέμα. Περνάμε τώρα σε δύο άλλα θέματα. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο όμως πια. Περνάμε στο σημείο 18. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μαρία Μπάντια Ικουτσέτ. Η μεταμόρφωση της Ευρώπης σε ένα κόσμο μετά την κρίση. Έχετε τον λόγο. δέκα λεπτά, όχι παραπάνω. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω είναι μια προσπάθεια σημαντική και δύσκολη ταυτόχρονα να επιτευχθεί. Ακριβώς πρόκειται για μια γνωμοδότηση, για μια έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας και για μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία συμβολική που αποκαλείται Ναυαρχίδα, Flagship Initiative. Νομίζω έτσι ακριβώς μεταφράζεται. Η Ναυαρχίδα της Στρατηγικής 2020. Και είναι σκόπιμο να ε, αποκαλούμε με αυτό το χαρακτηρισμό διότι η καινοτομία είναι ένας σημαντικός πυλώνας για την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για μας σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή όσον αφορά την παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και την επαγγελματική κατάρτιση φυσικά ακόμα. Στο σχέδιο που έχετε ήδη στα, ε, στους ε, χαρτοφύλακές σας βλέπετε ότι θέλουμε να υποστηριχθεί αυτή η καινοτομία, αυτή η πρωτοβουλία μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο που θα, θα εμπεριέχει όλες τις ε, ιδέες από τις αρχικές προτάσεις μέχρι τις τελικές τελευταίες όσον αφορά την καινοτομία στα θέματα νέων προτύπων ε, συναλλαγών και τη μέγιστο, το μέγιστο κέρδος που θα αποκομίζουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Εμένουμε και επιμένουμε στην ανάγκη να μεταμορφωθεί η Ευρώπη σε μια ζώνη βέλτιστων ακαδημαϊκών επιδόσεων, μεγαλύτερη κινητικότητα, επενδύσεις στην έρευνα, παράδειγμα όσον αφορά τις υποτροφίες Marie Curie. Σήμερα είχαμε και αναφορά σε αυτό το θέμα. Να πετύχουμε μια ζώνη έρευνας στην Ευρώπη και να μεγιστοποιήσουμε τις που προσφέρονται από το Ευρωπα... για το ευρωπαϊκό δυναμικό Έρευνα. Θέλουμε περισσότερη έρευνα στην Ευρώπη. Θέλουμε οι ερευνητέ μα να παραμένουν περισσότερο στην Ευρώπη, να μένουν στην Ευρώπη, να μην χρειάζεται να εγκαταλείψουν την Ευρώπη, να πάνε αλλού για να κάνουν το ερευνητικό του έργο. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Επίση, έχουμε συνδυασμένε προσπάθειε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση, περιφερειακό, τοπικό, κρατικό και ευρωπαϊκό, ώστε να πρικοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη συνεργασία, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι παραμέτρου και συνιστώσει για την παιδεία, εκπαίδευση και τα πολιτισμικά. Επίση, υπογραμμίζουμε τη σημασία αυτή τη καινοτομία στα κοινωνικά για να ανταποκριθούμε στι κοινωνικέ ανάγκε. Προποθέσει εργασία, όροι και προποθέσει βελτιωμένε για την εργασία. Επίση, για τα υγειονομικά και την υγεία, βελτίωση. Τονίζουμε επίση τη σημασία τη έρευνα, ιδιαίτερα στον τομέα των κοινωνικών επιστημών τον αγώνα, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες ε, όπως επιστήμη κατά της φτώχειας. Αυτά είναι σε αδρές γραμμές, αυτά που θέλουμε να πετύχουμε και προτείνουμε στην έκθεσή μας. Όπως γνωρίζετε πάντα, οι απόψεις, οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι πολύ σύντομες. Έχουμε πολύ περιορισμένο χώρο για να διατυπώσουμε απόψεις και θέσεις μας. Όποιος ενδιαφέρεται, συνιστώ να διαβάσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ θα ήθελε να τοποθετηθεί από αυτόν. Παρακαλώ εσείς, έχετε τον λόγο. Thank you very much. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Χαιρόμαστε πολύ που αυτή η Επιτροπή έχει δώσει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ήτρε, γιατί όπως βλέπετε στην ανακοίνωση της Κομισιόν ε, η καινοτομία θέλουμε να είναι εγκάρσια πολιτική των διαφορών πολιτικών της Ένωσης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υποστηρίζετε αυτή την γνωμοδότηση και η Κομισιόν συμμερίζεται τις απόψεις της ηγήτριας ότι θα πρέπει να ε, ξεπεράσουμε ε, ότι η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικά και είναι σημαντική η ποσότητα αλλά και η ποιότητα των πόρων ταυτόχρονα. Η Σιγήτρα επίση τόνισε τη σημασία τη δημιουργικότητα τη Ευρώπη, τη δημιουργικότητα στην έρευνα και σε άλλου τομεί και η Ένωση της Καινοτομίας θα ήθελε αυτές οι ιδέες που δημιουργούνται από ερευνητές, από καλλιτέχνε να αξιοποιηθούν, να φτάσουν στην αγορά και ε, στη τελευταία ανάλυση να δημιουργήσουν αύξηση και θέσεις απασχόλησης για την Ευρώπη σημασία της ε, υποστήριξης της υπεροχής στην έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως γνωρίζετε, η έρευνα στην Ευρωπαϊκή στηρίζεται στο κριτήριο υπεροχής και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα εις βάρος αυτού του κριτηρίου. Θα πρέπει να συμπληρώνει τα άλλα. Η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας είναι σημαντική. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας υπενθυμίζει για πρώτη φορά ε, ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χώρο, ευρωπαϊκό χώρο για την έρευνα και θα θέλαμε να συζητήσουμε ε, την πέμπτη ελευθερία, την ελευθερία των ε, ιδεών και των γνώσεων. Και η Κομισιόν συμμερίζεται την έκκληση που κάνετε στα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις πολιτικές μετά την έρευνα της μεγέθυνσης που έγινε από την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν τα εθνικά σχέδια και ε, προσυπογράφουμε αυτά που είπατε σχετικά με την σημασία της ενσωμάτησης, της ε, έρευνας, της κατάρτισης, της καινοτομίας στα σχέδια τους. λοιπόν, σας ευχαριστώ για την στήριξή σας και αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνει η Κομισιόν ε, προς την Επιτροπή αυτή, θα είναι χαρά μας να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και για την, την Επιτροπή. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της διάταξης. Και σχετικά γοργά πρέπει να προχωρήσουμε. Περνάμε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ευρυζωνικότητας και η κυρία Μπεναράμπα θα λάβει τον λόγο. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ε, ε, donc, le ε, πρέπει να επενδύσουμε στην ευρυζωνικότητα στην Ευρώπη και να επωφεληθούμε ε, από την έλευση της ψηφιακής ε, περίοδου. Είναι σημαντικό για το μέλλον των Ευρωπαίων και για τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο στόχος μας είναι η ευρυζωνικότητα να είναι σε διάθεση όλων των Ευρωπαίων μέχρι το 2013. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες πάνω από 30 Mbit το δευτερόλεπτο ε, μέχρι το 2020. Η ανάπτυξη της ευρείας ζώνης ε, δεν είναι αυτός σκοπός και δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των δημοσίων πολιτικών ε, βιώσιμης ανάπτυξης, ποικιλομορφίας, κοινωνικής ένταξης και πολιτιστικής ένταξης, αλλά θα πρέπει να συνεισφέρει. Ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι να τομίσουμε τη σημασία του περιεχομένου ποιότητας και των διακυβευομένων ε, της ευρυζωνικότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη γνώση. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα προάγουμε την ε, γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία, την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Θα υπάρξει πρόσβαση στον πολιτισμό και ανάπτυξη του διαπολιτιστικού διαλόγου. Ακριβώς γι' αυτό η γνωμοδότηση αυτή βασίζεται ε, σε προτεραιότητες όπως οικονομική δημόσια χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε ζώνες που έχουν χαμηλό πληθυσμό. Ε, η σύνδεση των δημοσίων υπηρεσιών, κυρίως των σχολείων, ε, με δίκτυα ευρεία ζώνης σε, όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η εκπαίδευση γενικά και η εκπαίδευση για τα ψηφιακά θέματα, η προώθηση του περιεχομένου ποιότητας και η προώθηση των πολιτιστικών εργαλείων. Με αυτόν τον τρόπο θα προάγουμε μια αλληλέγγυα κοινωνία ε, σεβόμενη τις ε, δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των προοπτικών ε, της Ευρώπης 2020. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα είναι η βάση της οικονομίας μας, του πολιτισμού μας, της κοινωνίας μας και με αυτόν τον τρόπο προάγουμε και την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν μπορώ... Ε, δεν ολοκλήρωσα την γνωμοδότησή μου. Περιμένω τα σχόλιά σας με ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα μου περάσετε ιδέες ούτως ώστε να καταλήξουμε σε, επικοδομητικές, σε μια επικοδομητική έκθεση. Ε, κυρία Φαχάιν, παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να προτείνω ίσως στο μέλλον με τους σκιώδεις εισηγητές να έχουμε εντονότερη ανταλλαγή απόψεων και να συνεχίσουμε για αυτό το σημείο όπως και με την κυρία Κάμεβε το πιο πριν όσον αφορά τις συχνότητες γιατί είναι σημαντικό οι πολιτισμικές πτυχές σε όλη την τεχνική συζήτηση για την ευρυζωνικότητα και τις συχνότητες να προαθούν τα πολιτισμικά. Είναι αρκετά δύσκολο αυτά τα θέματα να ενταχθούν στη γενικότερη συζήτηση γι' αυτό πρέπει και σε αυτό το πλαίσιο να ληφθούν υπόψη Χαίρομαι για την περαιτέρω διαμόρφωση της συζήτησης και ελπίζω ότι θα έχουμε μια εντονότερη συνεργασία ώστε αυτά να προαχθούν όπως πρέπει. Υποστηρίζω απόλυτα την σκέψη του ότι η εξέλιξη των ευρυζωνικών όχι μόνο στον χώρο της Υπέτρου αλλά και συνολικά έχει μια σημαντική πολιτισμική πτυχή, την πρόσβαση στις γνώσεις, την πρόσβαση στα πολιτισμικά, ουσιαστικά αυτά που πρέπει να είναι προϋπόθεση για κάθε πολίτη. Να υπάρχει ελεύθερη προσπελασιμότητα σε αυτό το μέσο για τους πολίτες και μέσω αυτών, αυτής της δυνατότητας όλων των νέων τεχνολογιών. Και είναι λιγότερο ευνοημένοι οι χώροι της Υπέθρου και με πολύ βραδείς ρυθμούς και με παλαιά τεχνολογία που έχει ξεπεραστεί. Υποστηρίζω απόλυτα το έτοιμά σας. Ξεκινώντας από το ότι η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι ένα δημόσιο, θα έλεγα, αντικείμενο δημόσιας προαγωγής και προώθησης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να βοηθήσουμε ένα σημαντικό πολιτισμικό αγαθό και δεν είναι κάποιο παιχνιδάκι αναψυχής το οποίο, κάνει το παρακολουθεί κάποιος, είναι πρόσβαση στη γνώση και στη σύγχρονη σύγχρονη επικοινωνία. Και γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε, πιστεύω, ελπίζω, καλή συνεργασία στο μέλλον για να προαχθεί αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος. Ε, ευχαριστώ για αυτές τις πτυχές που συζητήσαμε, τη διαθεσιμότητα της υψηλής ταχύτητας, ευρυζωνικότητα. Αν θέλει κανείς να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός στις επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλους τομείς όπως ε, τις ε, κοινωνικές επικοινωνίες. Ε, το συντομότερο θα επενδύσουμε και θα το κάνουμε διαθέσιμο στην Ευρώπη σε όλες τις περιοχές αστικές και αγροτικές, τόσο καλύτερη θα είναι η κοινωνία. Η ευρυζωνικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα για την επικοινωνία, και για, τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Αν δούμε την ιστορία του κόσμου, θα δούμε διάφορες εφευρέσεις που άλλαξαν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως η εφεύρεση του τροχού, της ατμομηχανής, του αυτοκινήτου και μέχρι την, τη σημερινή εποχή η ευρυζωνικότητα και η διαθεσιμότητα της ευρυζωνικότητας είναι αναγκαία σε όλη την Ευρώπη ε, αλλά αυτή τη στιγμή ε, ποικίλει σε ταχύτητα. Σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχει καθόλου. Το χρειαζόμαστε, έχει το δυναμικό να βοηθήσει κάθε περιοχή να αναπτυχθεί και θα αλλάξει τους παράγοντες που ε, θα αποφασίζουν ε, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες να εγκατασταθούν. Διότι με την σωστή ευρυζωνικότητα και τις πωλήσει μέσω του διαδικτύου οι τοποθεσίες των, των διαφόρων φορέων θα αλλάξουν. Ευχαριστούμε πολύ. Λόκεγκάτ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Επειδή τα πάω πολύ καλά στα δανέζικα σήμερα, θα μιλήσω και πάλι στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια πολύ καλή και σύντομη δήλωση. Ε, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κάπως ε, το θέμα. Εν μέρη θα συμφωνούσα με αυτά που έχουν ελεγχθεί. Μόνο εν μέρη όμως η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει εθνικά σχέδια βριζονικότητας και, αποτελε... και τους πίνακες με τα αποτελέσματα επίσης. Και σε ό,τι αφορά του πίνακε, ως αποτελεσματικό εργαλείο που έχει θετική επίδραση σε άλλους τομείς, αυτό το υποστηρίζω. Σε ό,τι αφορά τα, σχέδια, τα εθνικά σχέδια βριζονικότητας θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ε, μία πρόσβαση με βάση την αγορά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προτιμηθεί. Θα πρέπει να είμαστε επικριτικοί ως προς τη χρήση των δημοσίων ενισχύσεων. Ε, υπέβαλα κάποιες τροπολογίες εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού Υπάρχουν θετικές επιδράσεις ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές. Η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες να λαμβάνουν κάποιες υπηρεσίες και οι δυνατότητες ε, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Αυτά ήθελα να πω και προσβλέπω στη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση, Ραχάνα. Σύντομα και περιεκτικά. Όλοι γνωρίζουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιες προτάσεις βρίσκονται πίσω από το πακέτο αυτό και μπορούμε να υποστηρίξουμε από την πλευρά μας αυτό το εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω σε σχέση με την αρμόδια επί της ουσίας ε, ε, επιτροπή. Θα πρέπει και οι δικές μας πτυχές να ληφθούν υπόψη στο μέτρο του εφικτού από αυτήν. Διότι για έναν πάροχο ή για εκείνους που διαθέτουν συχνότητες στο διαδίκτυο δεν, πρέπει να, δεν είναι πάντα ενδιαφέρον και στην πιο απόμακρη περιφέρεια να επενδύσει. Εκτός αν έχουμε δορυφορική προσπελασιμότητα. Δύσκολα είναι προσπελάσιμα τα ε, πεδία, τα ε, εδάφη ε, των πιο απομακρυσμένων περιοχών χωρίς πρόσθετες επενδύσεις. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν είναι δυνατόν ένας γεωργός κάπου σε ένα απόμακρο μέρος να πληρώνει απίθανα ποσά, σύλληπτα ποσά για να έχει πρόσβαση. Δεν το κάνει αυτό. Θα πρέπει να ενδιαφερθούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα με βιώσιμο, προσιτό τρόπο. Φυσικά με την τιμολόγηση συναρτάται. Τώρα, όταν έχουμε εδώ δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020, θυμάμαι τι έλεγε αυτή η έκθεση, είναι μ, θαραλέο και ακούγεται και καλό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Η ευρυζωνικότητα είναι ένα μέσο ακριβώς. Οι πολίτες να διασυνδεθούν μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση σε γνώσεις που διαφορετικά δεν θα είχαν. Όλα αυτά είναι σαφή βέβαια, αλλά με την αναγκαία σύνεση και επιφύλαξη ότι όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν χωρίς να επιβαρυνθούν ή να ζημιωθούν κάποιοι άλλοι τρίτοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπόρις. Πολύ σύντομα. Μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά κλείνουμε. Ε, Ευχαριστώ. ευχαριστω διαφωνω με τον δανό συνάδελφο. Σήμερα μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Και αυτή αφορά και την ευρεία ζώνη. Σήμερα η Κεντρική και η Ανατολική Ευρώπη έχει μία ενίσχυση από τα Ταμεία Συνοχής για να αναπληρώσει την καθυστέρηση που έχει ε, καθυστέρηση δεκάδο, ε, δεκαετιών συγγνώμη, σε ό,τι αφορά την ευρεία ζώνη. Υπάρχει ένα πρόβλημα επενδύσεων που διαρκεί. Η τελευταία στιγμή, τη στιγμή που θα πρέπει να επενδύσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ένα δίκτυο ούτω ώστε τα μικρά χωριά και ο καθένας να έχει πρόσβαση ε, στην ευρεία ζώνη, αυτό είναι τεράστια σημασία. Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν τα κονδύλια των ταμείων συνοχή, ούτω ώστε να βοηθήσουμε και να προάγουμε και τι επενδύσει ε, στην ευρεία ζώνη. Να μην το ξεχνάμε αυτό και στι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ, γιατί είναι πάρα πολύ αποτελεσματικέ αυτέ οι επενδύσει και κεφαλαιόδου σημασία. Σα ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ τώρα. Ναι, Έχετε τον λόγο δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Η Κομισιόν θα συμφωνήσει σχεδόν με όλα τα σχόλια. Ένας από τους μείζονες σκοπούς είναι να φέρουμε την ευρεία ζώνη και στην Ήπεθρο. Είναι προτεραιότητα και έχουμε εξετάσει όχι μόνο την διασυνδεσιμότητα, όλη δηλαδή η Ευρώπη να έχει ευρεία ζώνη μέχρι το 2013, αλλά μέχρι το 2020 να υπάρχει ευρεία ζώνη, αλλά και με εύλογη ταχύτητα 30 Mbit σε όλους το δευτερόλεπτο. Ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ πόλεων και υπαίθρου, υπάρχουν διαφορές μεταξύ του κόστους, αλλά η στρατηγική μας εστιάζεται στην ε, ιδέα ευρεία ζώνη για όλους. Έγιναν σχόλια τώρα για τη χρήση των δημοσίων κονδυλίων και των δημοσίων ταμείων. Είπαμε ότι η προσέγγιση μας είναι μια προσέγγιση που να βασίζεται στην ε, αγορά. Η ευρεία ζώνη της επόμενης ε, γενιάς ε, θα είναι δαπανηρή και τα περισσότερα κονδύλια θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά θα υπάρξουν τομείς που δεν θα επενδύσουν, όπου δεν θα επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας. Εκεί ακριβώς υπησέρχεται ο δημόσιος τομέας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ρόλο του πολύ προσεκτικά, να παίξει το ρόλο του πολύ προσεκτικά. Το 2009 η Κομισιόν ε, εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τι τις κρατικές για την χρήση της ευρείας ζώνης. Συμφωνούμε με αυτά που είπαν οι περισσότεροι ομιλητές και ευχαριστούμε την ε, Επιτροπή σας για τη συνεισφορά της. Euh, Σύντομη, λακωνική. Υπόθηκαν πολλά πράγματα για την διαπραγμάτευση που γίνεται για τη γνωμοδότηση αυτή θα γίνει μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών πολύ σύντομα. Η σχέση με το φάσμα της ραδιοτηλεόρασης είναι πολύ σημαντικό. Το οικονομικό διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό επίσης. Το θέμα δεν είναι αμυγός τεχνικό, έτσι, είναι και οικονομικό. Αυτά έχω να πω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε στην ομάδα των σκιωδών και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Να υπενθυμίσω ότι στις 4 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, εκπνέει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Και κάτι άλλο, επίσης, να μην το ξεχάσουμε ότι... Τι είναι? Ναι. Και έχουμε το θέμα της μεταμόρφωσης Ευρώπης σε με, μετα, ε, περίοδο μετά της κρίσης και της κυρίας Μπαντία 2 Δευτέρα Φεβρουαρίου. Όλα δηλαδή την, την επόμενη εβδομάδα, εντάξει, σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται εδώ, κοντά μου, εδώ. Και περνάμε στο σημείο 20 τώρα. 20. Παρακαλώ κύριε Μπόρις. Σημείο 20. Έχετε κάτι να πείτε για το σημείο 20 εσείς. Το σημείο 20 είναι έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτές τις αποφάσεις. Δεν υπάρχει, όχι. 21. Διάφορα. Ο κύριος Μπόρις, παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Και με συγχωρείτε, θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσατε να αποστείλετε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ε, δυνατότητα χρήσης ε, των κονδυλίων για ε, το πρόγραμμα Εράσμους έτσι ώστε να βοηθήσουμε φοιτητές της Λευκορώσους. Θα ήθελα εδώ να δω, το, για το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο έχει να κάνει με μια αποστολή ερώτησης προς την Εκομισιόν κύριε Μπόρε, Θα μπορούσα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όλα αυτά είναι άτυπα. Μια επίσημη ερώτηση μπορείτε μέσω τη δική σα κοινοβουλευτική ομάδα να διατυπώσετε. Είτε μπορείτε να την να αποκοινούμε άλλου ευρωβουλευτέ να την κάνετε. Ή ο ίδιο μπορείτε γραπτό να υποβάλλετε ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κανόνε όμω και δεν μπορεί η Επιτροπή να του αγνοήσει. Το πρόγραμμα Έρασμό ε, έχει διευρυνθεί στι υποψήφίε προ ένταξη χώρε και τα κράτη των Βαλκανίων και την Τουρκία. Οι άλλε χώρε δεν έχουν ενταχθεί ακόμα. Μπορώ να σα πω από τον προπολογισμό του, Εράσμου, του Έρασμος δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά. Θα μπορούσαμε ώστε το έτοιμά σα να καλυφθεί να σκεφτούμε αν για τον εξωτερικό πολιτικό τομέα αν θα μπορούσαμε κάποια κονδύλια να χρησιμοποιήσουμε και να δοθεί μια τέτοια δυνατότητα. Τότε πρέπει να επιλεγούν κάποιε δράσει. Στου τομεί μα δεν γίνεται αυτό με κανένα τρόπο. Έχουμε κανόνε που πρέπει να σεβαστούμε και είναι σαφή τα όρια και έχουν καθοριστεί. Οι χώρε πρέπει να συμμετάσχουν αυτές οι χώρες και η Βοσνία και η Κροατία συμμετέχουν με τη βοήθεια των μέσων ΙΠΑ που τους καταβάλλονται αυτά τα κονδύλια. Και ξέρω ότι για αυτέ τι χώρε που το χρειάζονται και αυτέ πρέπει με άλλο τρόπο να προσπαθήσουμε να βρούμε μια δυνατότητα. Έχουμε και συζητήσει και ανταλλαγέ με την Κίνα. Γιατί δεν μπορεί κανεί με του γείτονέ μα να βρούμε μια νέα δυνατότητα. Αλλά αυτέ οι νέε δυνατότητε θα υπάρξουν γενικά, γενικόλογα με τα νέα προγράμματα ίσω. Τώρα όμως ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει κάπως αυτό το θέμα για κάποιους φοιτητέ ε, μέσω κάποιων κονδυλίων που στο πλαίσιο της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής θα μπορούσαν να διασφαλιστούν. Πρέπει να μεριμνήσουμε από κοινού. Ευχαριστώ για αυτό το έτοιμο. Κύριο κύριος Μιγκάλσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα αν επιτρέπετε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το οποίο διατύπωσε ο συνάδελφος κύριος Μπόρις. Σωστό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια που αναφέρατε και σε σχέση με την προφορική ερώτηση και τον συντονισμό όσον αφορά την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Εντάξει, όμως η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι πραγματικά δραματική. Οι φοιτητές βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και σε σχέση με τα όσα γίνονται σε σχέση με το Πανεπιστήμιο αρνούνται να ε, αποπέμψουν από το Πανεπιστήμιο ε, ε, φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις. Αυτό το συμμερίζονται και οι δημοκρατικοί πολίτε, οι δημοκρατικέ δυνάμει στη χώρα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου. Δεν έκαναν τίποτα, κανένα έγκλημα, επειδή συμμετείχαν σε μια διαδήλωση υπέρ τη δημοκρατία και τη ελευθερία και μέσω άτυπων διάβλων θα μπορούσατε ίσω να προωθήσετε αυτό το ερώτημα, αυτή την ερώτηση θα ήταν πραγματικά επικοδομητικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δοθεί απάντηση, έστω και άτυπα, αν γίνεται, και να δούμε μετά στη συνέχεια ποια συνέχεια θα δώσουμε, τι θα κάνουμε ω ξεχωριστή ερώτηση γι' αυτό. Η ημερομηνία επόμενη συνεδρίαση, 3η Μαρτίου, 9 11.30 το πρωί και 11.30 έως 12.30 και μετά 15.00 έως 18.30 το απόγευμα. Εντάξει, όλα εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους διερμηνείς. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Εντάξει, έκανα λάθος ολίσθημα, μετά δεν μιλάω σωστά τα αγγλικά, τα γερμανικά, κάνω λάθη. Εντάξει, τρομερό. Ευχαριστώ, γεια σας. You do not escape so easily.